Συνεχίζουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών και θα περάσουμε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ε, συνεδρίας της δικής μας Επιτροπής. Σημείο 2, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, παρακαλώ τα μέλη να ε, κοιτάξουν την ημερήσια διάταξη γιατί υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, για αλλαγές. Το σημείο 13 παραδείγματο χάρη έχει γίνει εισήγηση να αφαιρέσουμε τη μέση διάταξη στο σημείο 13. Η κυρία Γκουμάη είναι υπεύθυνη για το gender mainstreaming στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και αποφάσισε να μην υποβάλει τροπολογίες αυτή τη στιγμή. Οπότε το διαγράφουμε αυτό το σημείο. Το 14 τώρα, το σημείο της κυρίας ε, Ζαμπόρσκα, κατόπιν αιτήματος της Ιδίας, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση του σημείου αυτού μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Το 14, σημείο 14, αναβάλλεται η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση. Το σημείο 15 τώρα της κυρίας Γιάννα Κουδάκη. Επίσης κατόπιν ετοιματός της αναβάλλεται η συζήτησή του για την επόμενη συνεδρίαση. Συνοψίζοντας τα σημεία 13, το σημείο 13 μάλλον αφαιρείται και τα σημεία 14 και 15 αναβάλλονται για επόμενη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση του σχεδίου ημερησίας διατάξεως με αυτές τις αλλαγές. Σημείο 3 τώρα, ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχουμε δύο ακροάσεις, μάλλον δύο συνεδρίες διορθώνει η Πρόεδρος, για τις οποίες θα ήθελα να σας ενημερώσω. Ε, στις, ε, η συνεδρίαση αυριανή στις 30 Νοεμβρίου ε, που διοργανώνεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και έχει ως θέμα πώς να διευκολύνουμε τη ζωή των ευρωπαϊκών οικογενειών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα γίνει αυτό και προφανώς προσκαλούμε όλα τα μέλη σε αυτή την εκτακτή συνεδρίαση Επίσης ε, διεξάγεται ε, την 1η Δεκεμβρίου μια επίσημη ακρόαση από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30 που η επίσημη αυτή ακρόαση διοργανώνεται από την Επιτροπή Αλίας και το θέμα είναι γυναίκες και βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της αλίας. Προφανώς όλοι όσοι ενδιαφέρονται από τη δική μας Επιτροπή είναι προσκεκλημένοι. Σημείο 4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, έχετε στους φακέλους σας τα πρακτικά θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 5 της μερίσσιας διάταξης, δηλαδή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. είναι της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και ο αρμόδιος ηγετής είναι η κυρία Γιαόκα, Γιαρόκα, συγγνώμη. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λίβια Γιαρόκα λοιπόν για να μας παρουσιάσει την έκθεση και τις τροπολογίες και αύριο θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Κύριε Γιαρόκα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Thank Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είσαστε πραγματικά πάρα πολύ ευγενεί. Δεν θα χρησιμοποιήσω πολύ από τον χρόνο σα. Είναι μεγάλη η τιμή ω εισηγήτρια, μπορώ να προσφωνήσω, τα μέλη αυτή τη Επιτροπή, διότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή εργάστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τα δικαιώματα των γυναικών Ρωμά. Και η έκθεση ιδίας πρωτοβουλία ε, που αναφέρει σε αυτό το θέμα για μένα το να συντάξω τα συμπεράσματά μου όσον αφορά την έκθεση ήταν εύκολη υπόθεση με βάση αυτή την εμπειρία και τη γνώση σας. Τα σημεία τα οποία τις περισσότερες φορές προσπαθώ να εντάξω σε αυτή την έκθεση και έχοντας διαβάσει αυτή την έκθεση μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία για τα νομικά επιχειρήματα, για μια νομική βάση για στο ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη. Πολύ περισσότερο από την ε, περιγραφή του πώς θα έπρεπε το θεσμικό οικοδόμημα να ε, δημιουργηθεί στο τέλος και υπάρχουν και συστάσεις σχετικά. Πολύ λίγα μπορούν να ενταχθούν στο κείμενο από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Αυτό που θα ήταν όμως το πιο σημαντικό μήνυμα από τη δική μας ομάδα Ευρωβουλευτών και στη συνέχεια από το σύνολο του Ευρωκοινοβουλίου για αυτό το θέμα είναι τα πολύ αρνητικά ποσοστά ανεργίας των γυναικών Ρωμά. Υπό τον κομμουνισμό, κομμουνιστικό καθεστώς ε, είχαμε ε, μεγάλο ποσοστό που είχαν και ε, κάποιες ε, δυνατότητες. Τώρα όμως ε, μεγάλο ποσοστό αυτών των γυναικών είναι ευάλωτες, είναι άνεργες, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν να φάνε και σε σχέση και με τους άντρες βρίσκονται σε χειρότερη ακόμα μοίρα. Είδαμε ότι η αρνητική διακριτική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες δεν μπορεί να συγκριθεί πραγματικά στην αρνητική διακριτική μεταχείριση βάρος των ανδρών της ίδιας εθνοτικής κοινότητας των συγκάνων ή γυναικών γενικά. Αυτό που είδαμε λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχει πολλαπλασιαστής ε, της επίπτωσης αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης στις ζωές τους. Προτείνω με πέντε τροπολογίες στο κείμενο να ενταχθούν αυτά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η πρώτη αρνητικης διακριτικης μεταχειρισης στις ζωε τους προτεινω πεντε τροπολογιες στο κειμενο λόγο για ένα ισχυρό ε, για το θέμα της ανεργίας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας αυτών των γυναικών. Είδαμε και οι άντρες έχουν ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας και εκείνοι πλήττονται από πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας. Ακόμα βλέπουμε ότι ακόμα και αν οι άνδρες βρίσκονται εκτός αγοράς ε, εργασίας, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τη λειτουργία των οικογενειών λόγω αυτής της κατάστασης και πάντα οι γυναίκες και τα παιδιά είναι εκείνες που πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα εργασίας. Είναι πολύ πιο δύσκολο λοιπόν να καταφέρουν ε, οτιδήποτε. Αυτό βρήκανε οι ερευνητές ε, από την έρευνα επιτόπου. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν στρατηγική, ειδική, εξειδικευμένη, να βοηθηθούν οι γυναίκες ε, τσιγκάνες να μπορέσουν να βρουν εργασία, να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο διαφορετικά να διατηρηθούν αυτές οι οικογένειες των συγκάνων. Όλο και περισσότερα παιδιά ιδρυματοποιούνται για οικονομικούς λόγους, καταλήγουν σε άσυλα και ε, αναμορφωτήρια και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οικονομικά να μπορέσουν να αντέξουν και να επιβιώσουν αυτές οι οικογένειες. Ε, οι γυναίκες Ρωμά ε, όντας τέρισε κάθε επίπεδο όσον αφορά τις λήψεις απόφασης. Ε, αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει και με την δυνατότητα να βρουν δουλειά οι γυναίκες και να βρουν δυνατότητα να εκφράσουν τη φωνή τους, να αποκτήσουν δικαιώματα οι γυναίκες, οι τσιγκάνες. Και πιστεύουμε επίσης ότι στο τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, στο εθνικό επίπεδο και διεθνές επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Αυτές οι γυναίκες πρέπει να ενταχθούν. Δεν είναι μόνο οι αρμόδιες οι υπεύθυνε για τις οικογένειες. Θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικές μορφές στην κοινωνία, στον, στις μικρές κοινωνίες τις οποίες ζουν. Παραδείγματα έχουν δείξει ήδη ενώ υπάρχουν πολύ λίγες ε, τέτοιες γυναίκες ε, τέτοιες οργανώσεις ε, που να έχουν κάποια εξουσία, να έχουν κάποιο αξίωμα όταν έχουν ένα τέτοιο αξίωμα μπορούν να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές το επόμενο σημείο συνδέεται με εκείνο το οποίο ανέφερα το πόσα λίγα πράγματα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση για την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην έκθεση να βρούμε την ισότητα των φύλων, να αναγνωρίσουμε την ισότητα των φύλων ως τον κυριότερο στόχο. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ελπίζω το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη και την διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών σε σχέση με τους άντρες να την καταπολεμήσουμε. Το τελευταίο σημείο των προτάσεών μου αφορά το πώς τα στοιχεία τα οποία έχουμε για το φύλλο, για την κατάσταση για τις γυναίκες. Στην περίπτωση της στρατηγικής για τις γυναίκες Ρωμά θα έπρεπε να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις επιτυχίες ε, που έχουν, έχουμε σημειώσει ή και τις ε, αποτυχίες που έχουν σημειωθεί. Να γίνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους γνώμο, ε, δείκτες και στοιχεία για να αξιολογήσουμε τη στρατηγική και τα αποτελέσματά της. Είναι κάτι το οποίο έχει χρονική διάρκεια και πρέπει έτσι με τους δείκτες και τα στοιχεία να αντανακλάσουμε αυτά. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω αύριο τελευταίο αυτό. Γνωρίζω ότι σχεδόν όλοι από εσά ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα και για τέτοιου είδου έρευνες και επειδή έχουμε ζητήσει από πανεπιστημιακούς δύο εργάζονται μία στην Βουλγαρία που έχουν προσκληθεί και οι άλλοι 15 χρόνια έρευνας ε, έχει διεξαγάγει σε ιταλικά, ε, ε, σε ιταλικά στρατόπεδα θα έλεγα συγγνώμη σε καταβλισμούς τσιγκάνων ακριβώς και που έχει κάνει έρευνες σχετικά εκεί και αυτά θα ήταν στη διάθεσή σας αν μπορείτε να συμμετάσχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος της Επιτροπής σας ευχαριστούμε και για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για αύριο το απόγευμα. Φυσικά θα συμμετάσχουμε. Γνωρίζουμε τις ε, γνώσεις σας, γνωρίζουμε την προσήλωσή σας, την αφοσίωσή σας για αυτό το θέμα την ε, συμπόνια που έχετε για την τύχη και την κατάσταση των Ρωμά, για την ανεργία, την ε, έλλειψη εκπαίδευσης, ε, τα προβλήματα που έχουν και χαιρόμαστε όλος ιδιαιτερός που είσαστε αρμόδιοι για την εξέταση της κατάστασης των γυναικών και παιδιών Ρωμά. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα ήθελε το λόγο. Η κυρία Κορνέλισεν μας ζήτησε ήδη το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιαρόκα. Είναι μια πολύ καλή έκθεση αυτή. Είσαστε επαίων και αυτό πραγματικά αξίζει έχει και τους λόγους για τους οποίους θεωρείστε παίων και για τις τροπολογίες που μπορούν να υποστηριχθούν. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι λείπει θα ήταν πολύ σημαντικό πιστεύω να συμπεριληφθεί κάτι για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανταλλαγή καλών πρακτικών διότι αυτό που βρήκα συζητώντας αυτά τα θέματα και στην Ολλανδία όπου σε σχέση με τους Ρωμά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ειδικά προβλήματα η στερεότυπη εικόνα που ε, υπάρχει είναι ότι το να αναλυφθεί δράση δεν θα ωφελούσε. Τίποτα δεν θα άλλαζε τη θέση των συγκάνων ούτως ή άλλως λέγεται. Αυτό φυσικά είναι τεράστια ανοησία. Και υπάρχουν καλές βέλτιστες πρακτικές και πρέπει να διαδοθούν, να διαχυθούν ακόμα περισσότερο. Και πολλές καλές πρακτικές ε, που συναντούμε είναι σε δημοτικό επίπεδο. Οι Δήμοι και οι κοινότητε θα έπρεπε να προαθούν πολύ περισσότερο για την προαγωγική ανταλλαγή αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Θα ήταν εξαιρετικό αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, θα έλεγα. Και μια σύντομη ερώτηση για τη διαδικασία σε σχέση με αυτές τις τροπολογίες, διότι δεν κατάλαβα απόλυτα το τι θα γίνει είναι οι τροπολογίε αυτέ που θα καταθέσετε εσεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, στην ΛΥΜΠΕ, αλλά θα ψηφίσουμε και εμεί εδώ στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, υπάρχει ευκαιρία για μα, να εμπλακούμε, να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Ίσως επειδή έχασα τη συνάντηση των συντονιστών και δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορείτε να μας το αποσαφηνίσετε αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Πάιβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να δώσω ε, ευχαριστίες στην κυρία Γιαρόκα για τη δουλειά που έκανε για αυτήν την έκθεση αλλά και για τη δουλειά που έχει κάνει στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο παρουσιάζοντας και τονίζοντας την κατάσταση των τσιγκάνων. Θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφραστεί και οι Επίτροποι θα συμμετάσχουν σε μια ακρόαση στην Επιτροπή αυτή αυτής εβδομάδας θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για τη δουλειά που διεξάγεται, το έργο που καλύπτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το ίδιο το θέμα των συγκάνων. Ξέρουμε πόσο αρνητική και σοβαρή είναι η διακριτική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν με αρνητικό τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι περισσότεροι ζουν σε κατάσταση περιθωριοποίησης και σε μεγάλη φτώχεια. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ότι υιοθετήθηκε μια οδηγία να καταπολεμηθεί η αρνητική διακριτική μεταχείριση με βάση την εθνοτική προέλευση, πράγμα το οποίο καλύπτει και τους Τσιγκάνους. Πολλά έχουν γίνει για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των ατόμων και για τη συνειδητοποίηση σε σχέση με τις περιπτώσεις των θυμάτων η αξία αυτή τη νομοθεσία είναι μεγάλη. Μπορούμε να ε, συνεργαστούμε με τα σώματα και τι ε, υπηρεσίε για την ίση μεταχείριση. Ήδη το 2008 δημοσίευσε μία ανάλυση νομικών μέσων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δυνατοτήτων και των μηχανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που σε σχέση με τα κράτη-μέλη θα μπορούν να υποστηρίζουν τα, μέτρα για την ε, ένταξη, την ε, ένταξη των ρωματων των Τσιγκάνων. Πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη για να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η δουλειά. Τον Απρίλιο εφέτος είδαμε τι είχε επιτευχθεί αυτά τα δύο χρόνια. Και επίσης για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε μία ανακοίνωση όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και οικονομική ένταξη, επανένταξη των Τσιγκάνων τονίσαμε σε σχέση και με το 2008 πόσο σημαντικό είναι αυτό το πεδίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η προοπτική του φίλου. Η Λίβια Γιαρόκα όπως είπε, οι γυναίκες τσιγκάνες, τα κορίτσια τσιγκάνες αντιμετωπίζουν ειδική αρνητική μεταχείριση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή. Βλέπουμε ότι αντανακλάται και με το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας και στα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα οικιακής βίας, οικογενειακής βίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την προοπτική του φίλου στη δουλειά που κάνουμε για την ε, ε, ένταξη των ε, τσιγκάνων. Ιδιαίτερα για την ισότητα των φίλων Η στρατηγική που υιοθέτησε η Επιτροπή το Σεπτέμβριο, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει Πολλέ προτεραιότητε. Η πρώτη είναι η οικονομική ανεξαρτησία. Η οικονομική ανεξαρτησία είναι που δίνει στα άτομα, γυναίκες και άνδρες, την ευκαιρία να διαμορφώσουν ανεξάρτητα το μέλλον τους. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 έθεσε στόχους ε, για ποσοστό απασχόληση 75%. Για να προσεγγίσουμε έστω και πόρο αυτόν τον στόχο πρέπει να φτάσουν πολύ πιο κοντά στην αγορά εργασίας αυτές οι γυναίκες που βρίσκονται τόσο μακριά από αυτήν σήμερα. Γυναίκες, ε, ιδιαίτερα άτομα με ειδικέ ανάγκες ή αναπηρίες ε, πρέπει να ε, τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει έναν εσωτερικό μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσέξει ιδιαίτερα την χρήση που γίνεται από τα κράτη-μέλη των διαρθρωτικών και άλλων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ένταξη αυτή. Περισσότερα θα αναφέρουν οι επίτροποι αυτή την εβδομάδα στην ακρόαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ελπίζουμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση αυτών των στοιχείων κατά τα τέλη του έτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια ανακοίνωση που θα συμπεριλαμβάνει ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των ρωμάτων συγκάνων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ευκαιρίες που θα δίνονται ε, για να υπάρχει στοχοθέτηση για την κατάρτιση, εκπαίδευση, παιδεία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, θα στοχεύουν αυτά τα μέτρα ιδιαίτερα στις ε, ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως τους συγκάνους. Έτσι λοιπόν η δουλειά αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και της Λίβια Γιαρόκα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Πριν δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Γιαρόκα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για αυτή την ερώτηση που έθεσε η κυρία Κορνέλισεν. Οι συντονιστές της Επιτροπής μας τον Ιούνιο αποφάσισαν ότι δεν θα εκδώσουμε ίδια γνωμοδότηση αλλά ότι θα εγκρίναμε κάποιες τροπολογίες, οι οποίες κατευθείαν θα υποβάλαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε επίσημα πώς θα γίνει, ε, θα εγκρίνουμε τις τροπολογίες και ευθύ αμέσως ε, θα τις υποβάλουμε στην Επιτροπή Ελευθερίων ε, και στις αρχές Ιανουαρίου είναι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Αν πρόκειται να γίνει ψηφοφορία βεβαίως τον Φεβρουάριο. Ε, κύριε Γιαρόκα, θα θέλατε να σχολιάσετε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά το βρίσκω πολύ αναζωογονητικό αυτό και εκτιμώ όλα τα όσα είπατε και τη δουλειά στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε ως κέρδος από αυτό. Ελπίζω ότι με την ίδια προσέγγιση θα αντιμετωπιστεί αυτό το έγγραφο. Αν μου επιτρέπετε, ένα από τα πιο σημαντικά θεμελιώδη θέματα από τα πιο θεμελιώδη ουσία αυτής της έκθεσής μου, πέρα από το, τα οικονομικά επιχειρήματα για το ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται οι γυναίκες, οι Ρωμά, για να μπορούν να ε, είναι ανεξάρτητες και να διαμορφώσουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν, είναι ένα συμπέρασμα σε αυτό που για πολλούς είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να, μην, να, να μπορεί η οδηγία περί μη αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης να λειτουργήσει υπέρ των Ρωμά, των Συγκάνων. Και ελπίζω και πιστεύω και εγώ, όπως και συνάδελφοι, ότι αυτό θα είναι ο στόχο μα. Αυτό το θέμα των συγκάνων μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο αν η οδηγία για την ε, αντιμετώπιση, τη ρατσιστική αντιμετώπιση μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσει στην Ευρώπη για τις ίσες ευκαιρίες και πρέπει με πολύ σοβαρό τρόπο να πάρουμε το ρόλο μας για να ενημερώσουμε και να προαγάγουμε αυτά τα εξαιρετικά μέσα, αυτά τα εξαιρετικά εργαλεία που θα ανακουφίσουν αυτή την κατάσταση της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης των τσιγκάνων πανευρωπαϊκά. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν στο να διαδοθεί αυτό το μήνυμα με πιο ε, ηχηρό τρόπο διαζώσης θα πρέπει να εμπλακούν και να συμμετάσχουν. Αυτό θα ήθελα να προτείνω, να εμβαθύνουμε περισσότερο στο να δούμε πώς οι αρχές και τα σώματα σε εθνικό επίπεδο θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα τόπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιαρόκα. Αύριο θα ψηφίσουμε για, την, ε, για τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 6 το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βάσει του άρθρου 50 συνεργαστήκαμε για αυτό το θέμα με την Επιτροπή Απασχόλησης. Η κυρία Πλάμπ είναι η συγγήτρια από πλευρά της Επιτροπής μας και για την Επιτροπή Απασχόλησης η συγγήτρια είναι η κυρία Σιμ. Η φτώχεια και οι γυναίκες. Ε, ένα φαινόμενο που βλέπουμε ανά τον κόσμο, μία ε, αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο η φτώχεια στις γυναίκες και στον κόσμο γενικότερα αλλά και ειδικότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πλάμ για να μας παρουσιάσει το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Θέλω ευθύ εξ αρχής ε, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι είμαι η συγγήτρια για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο ε, πρέπει να εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους σας ε, για την υποστήριξη που μας ε, προσφέρατε στο να οργανώσουμε το Σεπτέμβρη μια δημόσια κρόση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Όσον αφορά τώρα την έκθεση, βεβαίως ε, πρέπει και έπρεπε να σεβαστώ τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν τούτου θέλω τώρα να σας παρουσιάσω κάποια σημεία κλειδί, καθοριστικά κατά την άποψή μου και είναι στοιχεία τα οποία ε, διαμορφώνουν ε, το πρόσωπο της φτώχειας ε, στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, η φτώχεια έχει τρεις διαστάσεις. Τις αποκαλούμενες διαστάσεις 3G από τα αγγλικά Geographic Generation και Gender στα αγγλικά γεωγραφική διάσταση ε, φύλου και γενιάς. Ε, τώρα λοιπόν τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα λιτότητας για να καταπολεμήσουν ε, ε, την χρηματοπιστωτική κρίση και κοινωνική κρίση. Ε, πρέπει λοιπόν να γίνουν εντελεχείς αναλύσεις ε, πριν ληφθούν μέτρα λιτότητας και βέβαια και να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Οι γυναίκες ε, τώρα είναι θύμα της αναδιάρθρωσης κυρίως στο δημόσιο τομέα. Είναι θύματα των περικοπών προϋπολογισμού, χάνουν τη δουλειά τους η κρίση επηρεάζει τους ηλικιωμένου ε, και τα άτομα με αναπηρία και γενικότερα όλες τις ευάλωτες ομάδες. Το τρίτο στοιχείο έχει σχέση με την ύφεση. Ε, οι επιπτώσεις της ύφασης ε, είναι πολύ πιο σημαντικές Κυρίω σε ευάλωτε ομάδε που αντιμετωπίζουν πολλά μειονεκτήματα. Εδώ αναφέρομαι στις ηλικιωμένε γυναίκες, ε, στις μετανάστριες ε, που ανήκουν σε εθνοτικέ μειονότητε, ε, στις ανήπαντρε μητέρε, στις γυναίκες σε αγροτικέ περιοχές και σε άλλες παρεμφερεί ομάδε. Στη δική μου την έκθεση εξετάζω το θέμα τη φτώχεια, τη γυναικεία φτώχειας σε διάφορου τομεί. Ο πρώτος έχει σχέση με το θηλυκό πρόσωπο της φτώχειας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ληφθούν ισχυρά μέτρα. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υιοθετήσει ένα χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτός ο χάρτης θα προκύψει μετά από διαβουλέψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να βελτιωθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Και βεβαίως τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου ε, στα προγράμματα, στα σχέδια που καταρτίζουν για την έξοδο από την ύφεση. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει σχέση με τις ε, πολιτικές εργασίες και την κοινωνική προστασία. Αυτά είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια των γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ότι η δική μας η Επιτροπή εργάζεται ε, σε ενισχυμένη μορφή συνεργασίας με την Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και η Επιτροπή Απασχόλησης ήδη ενέκρινε τη γνωμοδότηση για αυτήν την έκθεση. Το τρίτο στοιχείο έχει σχέση με την ε, συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής, κυρίως των γυναικών που ζουν στη φτώχεια ή είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της ε, φτώχειας. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να προάγουμε τη συμφιλίωση ανάμεσα στην ιδιωτική μας ζωή και την εργασία, ε, να προάγουμε τις δυνατότητες βρεφονιπιακών σταθμών, έχοντας υπόψη ότι η δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη Βαρκελόνη το 2002 ε, ισχύουν αυτές μέχρι το 2010 αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να φέρω έχει σχέση με τη φτώχεια ανάμεσα στις ε, ηλικιωμένες γυναίκες. Οφείλουμε να προσφέρουμε ικανοποιητική κοινωνική ασφάλεια ε, στις ηλικιωμένες γυναίκες αλλά και σε ε, άτομα της οικογένειάς τους που έχουν αναπηρία. Εδώ αναφέρομαι σε ηλικιωμένες γυναίκες, ε, ιδιαίτερα τις ε, χαμηλοσυνταξιούχους. Ένα άλλο θέμα αφορά την βία που ασκείται στις γυναίκες και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην ενδοοικογενειακή βία, τη φτώχεια και την εμπορία ανθρώπων. Επόμενο στοιχείο, κοινωνικός διάλογος και κοινωνία των πολιτών για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια των γυναικών. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό κοινωνικό διάλογο. Το έβδομο θέμα που θέλω να φέρω έχει σχέση με τις, ε, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο Διαρθρωτικό Ταμείο και κυρίως ε, στο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο. Αναφέρομαι επίσης σε συγκεκριμένα προγράμματα ε, στο πλαίσιο της ε, συγχρηματοδότησης έτσι ώστε να υπάρχει ενεργός συμπερίληψη των γυναικών στην αγορά εργασίας και εξειδικευμένη κατάρτιση για να αποκτήσουν αυτές ε, τα ειδικά προσόντα που είναι απαραίτητα ε, για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης που θα προκύψουν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Βεβαίως εγώ είμαι ανοιχτή και μπορώ κάλλιστα ε, να συνεργαστώ ε, και να συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Περιμένω τις δικές σας τις απόψεις και τροπολογίες και θέλω επίσης να αναφέρω ότι το να λάβει κανείς, ε, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι εγώ σεβάστηκα τη διαδικασία και εγώ έχω πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι προσβλέπω ε, στα σχόλιά σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πλάμπ. Τώρα θα γίνει συζήτηση. Η κυρία Κρεντίνσκα έχει ζητήσει πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εξ ονόματος των συναδέλφων σίγουρα από πλευράς ε, του ΕΛΚΑ να, του, των εισηγητών σχεδόν εισηγητών να αναφερθώ σε αυτό. Θα μπορούσα λοιπόν να συνεχίσω στα αγγλικά λέγοντας ότι έχοντας ταυτοποιήσει στη στρατηγική 2020 μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της φτώχειας που δημιουργεί, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα στα θέματα φύλου, υπό το φως της ε, σημερινής οικονομικής, ε, χρηματοοικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Και η γυναίκα ως άτομο ε, εκτίθεται σε μεγαλύτερους κινδύνους ε, κοινωνικού αποκλεισμού και γι' αυτό είναι καθήκον για μας να παρεμβαίνουμε μέσω στρατηγικών και προγραμμάτων στην έκθεση αυτή και για τα διάφορα ε, πεδία ενδιαφέροντος δίνεται μια ανάλυση του γυναικείου προσώπου της φτώχειας. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όμως εξετάζοντας διάφορα θέματα διασφαλίζοντας την δίκαιη μεταχείριση, πρόσβαση σε ε, υγειονομική περίθαρψη, χωρίς διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την κοινωνική τάξη, ε, εθνοτική προέλευση, να ε, αναζητήσουμε την δυνατότητα να μπορέσει να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία στις ε, γυναίκες ε, δίνοντας δυνατότητα νομικής ε, υποστήριξης στις γυναίκες όσον αφορά και θέματα που αφορούν τους συζύγους τους ή τους πατέρες των παιδιών τους. Όλα αυτά θα πρέπει συνολικά να εξεταστούν σε σχέση με την, το, τη χάρτα των δικαιωμάτων των γυναικών. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι άνδρες. Δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους πατέρες, τους αδερφούς ή τους γιους. Πρέπει να έχουν οι γυναίκες πραγματικά δίκαιη μεταχείριση και να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για την Ευρώπη αυτά. Και με την προοπτική του φίλου πρέπει να είναι σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών και να αναγνωρίζονται από τις χώρες και με μαθήματα που θα μπορούν να υποστηρίζουν αυτή την ε, ε, συνιστόσα, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα να υποστηριχθούν οι γυναίκες. Και είμαστε εκείνες που πληρώνουν το αντίτιμο για την ε, ανάκαμψη όσον αφορά και την οικονομία χωρίς να είμαστε εμείς οι επικεφαλείς πληρώνουμε το αντίτιμο και στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία και βλέπουμε ότι η μάχη που δίνουμε για τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας στις ε, χώρες μας και στα διάφορα επίπεδα βλέπουμε ότι ολόκληρη ε, ε, πάρα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να, όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, να μπορούν να, καλύπτονται και οι ανάγκες των γυναικών. Πρέπει να υποστηρίξουμε οικονομικά τα ε, θύματα, τις γυναίκες ε, όσον αφορά την ε, απομόνωση, τον αποκλεισμό και τη φτώχεια. Πρέπει να υπάρξουν δίκτες που θα μπορούν να καλύπτουν αυτές τις πτυχές σε σχέση με τις γυναίκες. Πρέπει να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα, όπως δημιουργήσαμε ένα τηλέφωνο, έναν αριθμό τηλεφώνου για να ανταποκρινόμαστε στις ε, ε, κλήσεις ε, των ατόμων που έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν, να μπορέσουν να γνωρίζουν ποιο είναι και το πιο κοντινό νοσοκομείο, πώς μπορεί να υποστηριχθούν και να τύχουν ιατρικής περίθαλψης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορούν οι γυναίκες και να μπορούν να εργάζονται και να αντιμετωπίζουμε την περίπτωση ασθένειάς τους ή την εγκυμοσύνη τους να μπορέσουν σε κρίσιμες στιγμές σαν αυτές να μπορέσουν να υποστηριχθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μάισνερ τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, yes. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδη εισηγητρία για τους φιλεύθερους ε, και ε, τώρα λαμβάνω το λόγο εκ μέρους ε, της κυρίας Αντώνιο Παρβάροβα που είναι σκιώδη εισηγητρία εδώ στην Επιτροπή Γυναικών. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτά που μου έγραψε. Επειδή Μάλλον, ω δεύτερη σκιώδη συγγήτρια για την έκθεση αυτή, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά τη ε, που παρουσιάζει γενικότερα ε, σε ευρύτερο πλαίσιο το θέμα τη ε, γυναικεία φτώχεια, του θηλυκού προσώπου τη φτώχεια. Πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκε εργασία, να υπάρξουν πακέτα και άλλοι μηχανισμοί για κάθε μία ευάλωτη γυναίκα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών και να εξεταστεί, αντιμετωπιστεί η ζωή των γυναικών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι αυτό το πλαίσιο πολιτικής οφείλει να υπογραμμίσει ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι αρχές της Ευρώπης, οι νόμοι της για την ισότητα, ε, την κατάργηση διακριτικών μεταχειρήσεων έτσι ώστε να βελτιωθεί και η οικονομική κατάσταση των γυναικών. Αυτά έγραψε η συναδελφός μου και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Ε, πιστεύω ότι αυτά για τα οποία συζητήσατε στην έκθεση αυτή είναι πολύ καλά. Αναφέρατε ε, το θηλυκό πρόσωπο της φτώχειας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρει κανείς αυτό γιατί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη φτώχεια ανάμεσα στις γυναίκες από ότι ανάμεσα στους άντρες. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά κυρίως τις γυναίκες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που ε, συντάσσει έκθεση η Επιτροπή Γυναικών. Αυτό είχα να προσθέσω. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Η Αντιπρόεδρος, κυρία Μωρή θα πάρει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι το εξής ε, και νομίζω ότι η συνάδελφος Πλάμ το γνωρίζει, αλλά είναι καθήκον που έχουμε εδώ στην Επιτροπή Γυναικών να μεριμνήσουμε ώστε να σταματήσουμε να εκριζώσουμε τη φτώχεια των γυναικών γιατί όσο αυξάνεται η φτώχεια τόσο περισσότερο πλέονται οι γυναίκες. Και η αύξηση του φαινομένου της φτώχειας έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις και επ' αυτού θα πρέπει να επικεντρωθεί η δράση μας. οι γυναίκες απασχολούνται με συμβάσεις ε, περιορισμένης ε, διάρκειας, κατέχουν ε, επισφαλείς θέσεις εργασίας και δεν μπορούμε απλώς να επιχαίρουμε διότι υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση για τις γυναίκες πλέον στην αγορά εργασία, γιατί αυτό ισοδυναμεί με επισφαλείς θέσεις εργασίας όπως σας είπα, και με συμβάσει προσωρινή διάρκεια. Ε, και άρα πλησιάζουν περισσότερο τη φτώχεια παρότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα ως προς τη θέση που κατέχουν αντίστοιχα οι άντρες και οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε μια λύση. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την επόμενη δεκαετία θα σημειωθούν, όπως δείχνουν εξάλλου και οι μελέτες, απώλειες της τάξης του 15% για τις θέσεις εργασίας με χαμηλή δίκευση. Αντίθετα, θα σημειωθεί αύξηση 15% των θέσεων εργασίας για τις ε, θέσεις υψηλής ειδίκευσης, αλλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση ε, γιατί αν δεν αναλάβουμε τα μέτρα που πρέπει, όπως μέσα στην έκθεση που σήμερα συζητούμε η κυρία Πλάμ, ξέρουμε ότι αυτό το 15% των θέσεων εργασίας που θα εκλείψουν, θα πλήξουν και πάλι τις γυναίκες. και οι γυναίκες θα είναι τα θύματα αυτής της απώλειας θέσεων ε, εργασίας ε, για ε, δουλειές χαμηλής ειδίκευσης. Δεύτερον, πάλι στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και ως προς την αύξηση των δεξιοτήτων, θέμα που μόλις τώρα σχολίασα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό την αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση, τη συνεχή εκπαίδευση αν βασιστούμε στην βασική εκπαίδευση ώστε να είναι καλύτερα και περισσότερο επιμορφωμένες οι γυναίκες τους ώστε να έχουν καλύτερη τύχη στην αγορά εργασίας αλλά αν αυτό δεν συνδυαστεί με αντίστοιχα μέτρα για την ε, συμφιλίωση οικογενειακής και τη ιδιωτικής ζωής τότε δεν θα ευοδοθούν οι προσπάθειές μας γιατί τα πτυχία των γυναικών δεν μπορούν να μετατραπούν σε θέσεις απασχόλησης. Αν βασιστούμε τώρα στη διαβίου μάθηση, στη συνεχή επιμόρφωση, ε, θα περιμένουμε από τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν τρεις ημέρες εργασίας, δηλαδή την κανονική δουλειά τους, ε, τη δουλειά που έχουν στο σπίτι και τη συνεχή επιμόρφωση. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να αναλυθούν μέτρα ούτω ώστε να είναι πιο ευέλικτα τώρα εργασία ε, για τις γυναίκες για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη διαβίου μάθηση για την πιστοποίηση ε, των δεξιοτήτων τους ούτω ώστε ισότιμα να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια οι γυναίκες. Αλλιώς θα έχουμε πολύ δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και θα ε, αποκλείσουμε τις γυναίκες μέσα στη φτώχεια. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σέσκοβα τώρα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμμετείχα στην άματος και θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Ίσως ε, αυτά που θα πω να μοιάζουν με αυτά που είπα ε, στην Ακρόση. Εγώ προέρχομαι από την Τσεχία. Εκεί λοιπόν το 9% του πληθυσμού ζει στη φτώχεια. Αυτός ο αριθμός ε, μοιάζει μικρός σε σχέση ε, με τους ε, υπόλοιπους αριθμούς που σχήνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα να φέρω άλλα στατιστικά δεδομένα, αλλά θέλω να σας πω ότι όσον αφορά την Τσεχία έχουμε μονογονοϊκές οικογένειες, ε, γυναίκες χωρίς σύντροφο, με μικρά παιδιά Αυτές λοιπόν ε, δεν μπορούν να εργαστούν εύκολα στην αγορά εργασίας, δεν βρίσκουν δουλειά και απειλούνται από τη φτώχεια. Ε, στην Τσεχία ε, έχουμε λοιπόν μονογονικές οικογένειες όπως σας είπα και από αυτές τις οικογένειες το 90% εκπαιδεύονται και αναθρέφονται από ε, τις γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές, όπως σας είπα, δεν μπορούν να εργαστούν εύκολα και πιστεύω ε, το γεγονός αυτό οδηγεί στο ότι οι γυναίκες αυτές είναι φτωχές και δεν μπορούν εύκολα να οργανώσουν βοήθεια για τα παιδιά. Αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες ε, στο να βρουν ε, ευέλικτο ωράριο εργασίας και έχουν και δυσκολίες ε, και όσον αφορά στις ευέλικτες συμβάσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για αυτές τις γυναίκες είναι καλό να υπάρχουν σταθερά ωράρια εργασίας Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει έλλειψη κενών θέσεων στους, ε, στα νηπιαγωγεία στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ε, πράγμα που πρέπει να εφίσταται για να μπορούν να εργαστούν οι γυναίκες αυτές. Πολλές από αυτές τις γυναίκες επιθυμούν να εργαστούν και δεν θέλουν να εξαρτώνται από το κοινωνικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες. Πιστεύω ότι οι γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά και οι οποίες κατά την άποψή μου φύγονται από τη φτώχεια ε, οι μητέρες αυτές είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν ε, στις απαιτήσεις της ζωής. Ε, πολλές εξ αυτών δεν έχουν και διατροφή από τον πρώην σύζυγο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιο ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τώρα λοιπόν, μιλώντας για επισφαλείς θέσεις εργασίας, δεν σκεπτόμαστε άραγε ότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι τις συμβάσεις εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λεωτάρ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια γιατί κατόρθωσε να πραγματευτεί μία σειρά σημείων που πραγματικά οδηγούν τις γυναίκες ε, στη φτώχεια. Έθεσε το δάκτυλο επί του τύπου των ύλων, επί των τύπων των ύλων, για να είμαι πιο ακριβής, μέσα στην έκθεση και θα την υποστηρίξουμε. Θα ήθελα να επιμείνω για τη σημασία ενός ζητήματος που αναφέρετε και εσείς μέσα στην έκθεσή σας και δηλώνω ικανοποιημένη. Λοιπόν, πρόκειται για τη φτώχεια των πιο ηλικιωμένων γυναικών που είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη και συχνά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα η κρίση για να γίνουν εξοικονομήσεις ε, στα ασφαλιστικά συστήματα, τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εφ' εξής σε εκθέσεις μας, ότι αυτό συνιστά μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια, κυρίως στις πιο ηλικιωμένες ε, γυναίκες. Όταν λέμε ότι θέλουμε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αυτές οι γυναίκες, ε, λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να επιμείνουμε ώστε ε, να υπάρξει μια συνειδητοποίηση τη ε, διακριτική ε, μεταχείριση που υφίστανται οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι στην αγορά εργασία. Ε, δεν είναι λήψη βουλησή του που δεν συμμετέχουν. Πρόκειται για ένα πολιτισμικό φαινόμενο και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Και σα παραπέμπω και στην πράσινη βίβλο για τι συντάξει. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτή την έκθεση και τη θέση τη επιτροπή μα για αυτή την πράσινη βίβλο για τα συνταξιοδοτικά συστήματα που αναμένεται να συζητήσουμε τους προσεχείς μήνες. Είδου και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Περέσκιβας. Παρακαλώ. Κυρία Παρασκευά, ίσω δεν ξέρουμε αν πρόφερε σωστά η πρόεδρο το όνομα τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν παρίσταται κανεί ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπω κάποιο άλλο από πλευρά τη Επιτροπή θέλει αργότερα το λόγο. Ο κύριο Σιμάνσκι πάντω έχει εγγραφεί στον κατάλογο μιλητών. Παρακαλώ. Pani Przewodnicząca, Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να υποβάλω ένα ερώτημα, όπως και οι προαλήσαντες, ε, που αφορά στις μονογονοϊκές οικογένειες, αντρίπανδρες μητέρες. τίθεται το ερώτημα το θέμα της διατροφής που πρέπει να καταβάλουν οι ε, πρώην σύζυγοι στις ε, γυναίκες τους. Ε, το αποφεύγουν αυτό οι πρώην σύζυγοι. Κατοπίν ότι τα κράτη δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τεράστια βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω στην έκθεση αυτή να δοθεί σημασία στο ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν τα συστήματα οι ε, γονείς, ε, οι γονείς λοιπόν απεκδίονται των ευθυνών τους όταν ο πατέρας εργάζεται ε, εργάζεται και δίνει τα χρήματα στη νέα του οικογένεια και όχι στην προηγούμενη, στα παιδιά από την προηγούμενη. Αυτό λοιπόν είναι κρίμα. Οι γυναίκες πολύ συχνά γνωρίζουν που εργάζεται ο πρώην σύζυγος αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν διατροφή. Πολύ συχνά οι σύζυγοι εργάζονται σε άλλο κράτος οι πρώην σύζυγοι. Αλλού είναι ο πρώην σύζυγος ε, και αλλού η μητέρα με το παιδί που ζουν σε μεγάλη φτώχεια. Εδώ λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμός, να υπάρχουν ε, συστήματα ενημέρωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον και ήθελα να το υπογραμμίσω γιατί σχετίζεται άμεσα με αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόσκα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές το θέμα της έκθεσης, διότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία συνέταξε έκθεση που ενέκρινε η παρούσα Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με θέμα ε, γυναίκα, γυναίκες και η φτώχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν η πρώτη σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Είπαμε ότι οι διαζεγμένες γυναίκες, οι μονογονικές ε, οικογένειες την να πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια. Το ίδιο ισχύει και για τις πιο ηλικιωμένε γυναίκες. Εγώ πιστεύω ότι και για τις δύο αυτές πληθυσμιακές ομάδες οι γυναίκες έχουν βυθιστεί στη φτώχεια και ε, ζουν σε αυτή τη δεινή κατάσταση διότι η κοινωνία δεν έχει αναγνωρίσει την αξία της μητρότητα. Δεν αναγνώρισαν την αξία της προσφοράς τους προς την κοινωνία. Συχνά οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες έχουν αναθρέψει πολλά παιδιά που εργάζονται, που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, αλλά οι ίδιες οι γυναίκες δεν ήταν σε θέση να εργαστούν για ε, μεγάλο αριθμό ετών και έτσι δεν έχουν κατοχυρωμένη σύνταξη και εξού και ένας αυξημένος κίνδυνος να βυθιστούν στη φτώχεια. Λοιπόν, ε, οι διαζεγμένες ε, τώρα γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα δίλημα. Τι να κάνουν, να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας ή να δεχτούν κυρίως τώρα που βιώνουμε και την κρίση θέσεις απασχόλησης με χαμηλότερη αμοιβή ε, και φυσικά που ζητούν χαμηλότερη ειδίκευση για να αναθρέψουν τα παιδιά τους γιατί συχνά δεν υπάρχει κανένας άλλος για να αναλάβει τα παιδιά. Πιστεύω ότι αν είχαν μεγαλύτερη υποστήριξη οι μητέρες δεν θα χρειαζόταν, δεν θα αναγκαζόντουσαν να δέχονται δουλειές μη αξιοπρεπείς, χαμηλά αμοιβόμενες, χαμηλής ειδίκευσης. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ε, το εξής. Για να είναι πολύ ε, αξιέπαινε προσπάθειες που κάνουμε για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκε. Αλλά ε, προσοχή, το μπορεί να, παρόλα αυτά να ζουν μέσα στη φτώχεια παρότι εργάζονται, διότι έχουν τέτοιες θέσει απασχόλησης, ε, χαμηλά αμοιβόμενε, έχουν παιδιά και οι ίδιες και τα παιδιά τους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας παρότι εργάζεται η γυναίκα. Γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ε, εχέγγυο η θέση εργασίας ε, κατά της φτώχειας. Ε, πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα μέτρα. Το εισόδημα πρέπει να είναι επαρκές για τα προστοζήν της οικογένειας. Στην κοινωνία μας έχουμε άντρες ε, και γυναίκες. Ε, έχουμε ζωντανά παραδείγματα που έχουν εργαστεί στο παρελθόν και ήταν τόσο χαμηλά τα εισοδήματά που αντιμετωπίζουν ε, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά και σας ευχαριστώ και συγχαίρω για πάλι την εισηγήτρια. Η Πρόεδρος, μάλιστα, σας ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόσκα. Τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Πάικ θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, Επιτροπής, εγώ είμαι από την ε, ε, διεθνή Περιποιότητας ή Ισότητας των Δύο Φύλων, το ίδιο και μου και ευχαριστώ την εισηγήτρια που μας υπέβαλε την έκθεσή Πράγματι η φτώχεια έχει κυρίως θελικό πρόσωπο και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι γυναίκες υποφέρουν κατά κύριο λόγο στην στρατηγική για την ισότητα των δύο φίλων όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε υπογραμμίσει αυτό το σημείο, κυρίως όσον αφορά την οικονομική αυτάρκεια. Και επισημαίνουμε το ότι οι άντρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Επίσης, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος όπως και της διαφοράς στο μισθολογικό προτείνουμε ε, το ότι ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις συμβάσεις εργασίας γιατί μερικές φορές αυτές εντείνουν το μισθολογικό χάσμα. Ο, η συγκήτρια και άλλοι μίλησαν για την στατική του 2020, μίλησαν για το στόχο ε, μείωσης της ε, φτώχειας, ε, ε την ε, πρωτοβουλία Ναυαρχίδα που θα έχει σχέση με το θηλυκό πρόσωπο της φτώχειας. Δεν λέμε ότι δεν θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια γενικότερα, αλλά θα πρέπει να ε, εξετάσουμε κυρίως τη διάσταση του φύλου στον τομέα αυτό. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι κάποια διαφωνία που έχω εκεί που ε, μιλάτε για τον χάρτη, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Γυναικών. Νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Γνωρίζω ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν έναν τέτοιο χάρτη. Ο χάρτης αυτός ε, έγινε η βάση της στρατηγικής μας και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστούν ε, τα ίδια δικαιώματα, ε, και να ενισχυθούν τα δικαιώματα αυτά, κυρίως ε, αναφέρομαι εδώ στην οδηγία περί άδεια μητρότητας. Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στο αρμόδιο Συμβούλιο. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν θεωρεί ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρχει χάρτης, ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων γυναικών. Αυτό ήθελα μόνο να υπογραμμίσω και κατά τα άλλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Πλάμ τώρα θα κάνει τις καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ε, άκουσα ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και προσοχή και την παρέμβαση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους. Θα λάβω υπόψη τις θέσεις σας. Όταν συζητούμε για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως λέω μέσα στην έκθεση, φυσικά μιλάμε και για τις μονογονικές οικογένειες και θα το λάβω υπόψη στην έκθεσή μου. Νομίζω πρέπει επίσης να προσθέσουμε μια κατηγορία, τις μετανάστριες από διάφορα εθνοτικά υπόβαθρα διότι μιλήσαμε και για την έκθεση της κυρίας Γιάρλακα για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των γυναικών ε, Ρωμά. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλές διαστάσεις ε, που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση για την απασχόληση και το είδος των εργασιακών συμβάσεων που συνήθως προσπογράφουν οι γυναίκες. Ε, προφανώς ε, ε, μπορεί αυτό να επηρεάζει και επηρεάζει τα ασφαλιστικά συστήματα. Κάποιος μας μίλησε για τις άδειες μητρότητος. Σε κάποια κράτη-μέλη η μητρότητα τιμωρείται σε εισαγωγικά και αυτό επηρεάζει αρνητικά τα ασφαλιστικά συστήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στη Ρουμανία. Το 85% των πληρωμών ε, για μία άδεια μητρότητας επηρεάζει κατά 7% την σύνταξη που θα λάβουν αυτές οι γυναίκες στη συνέχεια κατόπιν. Ε, ο χάρτης, ο ευρωπαϊκός χάρτης για τα γυναικεία δικαιώματα, το τελευταίο σημείο δηλαδή που αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα ως ερετός αντιπρόσωπος να εκπροσωπήσω σωστά τους πολίτες μας και να ζητήσουμε ο χάρτης αυτός να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στην Επιτροπή και του Κοινοβουλίου γιατί ε, νομίζω ότι με αυτή τη συνεργασία θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όπερ και θα είναι υποφελές για τους πολίτες ε, της Ένωσης και το αναφέρω μέσα στην έκθεση γιατί με, μου είναι ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα αγαπητό. Ε, και είναι κομμάτι του συνολικότερου νομοθετικού πακέτου. Αυτό ισχύει και για τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να προαγάγουμε ε, ενεργά μέτρα, ούτως ώστε, όπως ε, σωστά είπε η κυρία Μωράνε, να σταματήσουμε να μειώσουμε τη φτώχεια που πλήττει τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ όλους πολύ και αναμένω τις τροπολογίες σας Προφανώς θα ξανασυζητήσουμε το θέμα και ευελπιστώ ότι μετά τις συζητήσεις ε, θα καταλήξουμε σε μια ε, πολύ καλή έκθεση, ε, εποφελής για τους πολίτες και χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Πλάμπ στις 9 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η καταληκτική μας ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών ε, και στις 26-27 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει το θέμα το Μάρτιο από την Ολομέλεια. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως σε αυτό το θέμα. Επόμενο σημείο πριν όμω ε, περάσουμε στο επόμενο σημείο θα παραχωρήσω την Προεδρία στην κυρία Μωρίνε, στην Αντιπρόεδρό μας. Ε, παρακαλώ. Euh, Σας ευχαριστώ. Προτείνω τώρα να εξετάσουμε το σημείο 7 για το σχέδιο έκθεσης ε, περί των προτεραιοτήτων και των γενικών χαρακτηριστικών ενός νέου πλαισίου πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αντιστρέψαμε τις θέσεις μας και τους ρόλους μας με την Εύα Μπρίτ Σφένσεν, διότι είναι η συγγήτριά μας για αυτό το θέμα. Ε, και μου ζήτησε η κυρία Μπρίτ Σφένσεν να προεδρεύσω αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ασκήσει πλήρως το ρόλο της συγγήτριας για το θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε λοιπόν το σχέδιο στις 14 Ιουλίου. Να σας θυμίσω ότι στη συνεδρίασή τους οι συντονιστές ζήτησαν άδεια για τη σύνταξη έκθεσης ιδίας πρωτοβουλία σχετικά με τις προτεραιότητες για τον προσδιορισμό ενός νέου πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το Μάιο του 2011 στα πλαίσια του πακέτου θύματα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα, μια στρατηγική, ένα σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εντάξουμε την ε, έκθεσή μας αυτό το σχέδιο δράσης. Επίσης, η σημερινή μας συζήτηση εγγράφεται σε, στο γενικότερο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την καταπολέμηση της, ε, γυναίκα, της ε, βίας κατά των ε, γυναικών που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Εύα θα Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσής σας, παρακαλούμε. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απόφαση που έλεβε να συντάξουμε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία σχετικά με τις προτεραιότητες και τον προσδιορισμό ενός νέου πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας και των γυναικών. Ε, είμαι λοιπόν η για αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι στην καρδιά του ζητήματος της ισότητας. Ε, σε μια κοινωνία όπου ε, ζουν υπό απειλή οι γυναίκες, υπό απειλή διώξεων, υπό απειλή βία, σε μια κοινωνία τέτοια ε, είναι ανέφικτο να ζήσουν οι γυναίκες. Πρέπει οπωσδήποτε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίσα δικαιώματα. Είναι υψής της σημασίας να πραγματευτούμε αυτό το ζήτημα. Ε, είμαι δε πλήρως πεπισμένη ότι υπάρχει σοβαρότατη δέσμευση από πλευράς ε, των μελών της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό με τρόπο ώστε από κοινού και με ουσιαστικό τρόπο να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτές τις ε, βιοπραγίες, σε αυτές τις βάναυσες πρακτικές. Είμαι αισιόδοξη βέβαια, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από κοινού και θα σας το αποδείξω ε, το Κοινοβούλιο το 2009 έκρινε ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση της ε, βίας κατά των γυναικών. Είχαμε επίσης γραπτή δήλωση το 2009 σε συνεργασία με την UNIFAM που επίσης, ε, όπου επίσης τα σώματα κατά της βίας, ε, κατά των γυναικών, το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, επίσης εργάζεται για αυτό το θέμα, διάφορα ψηφίσματα και συμβάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή δε στο σχέδιο δράσης για το 2010-2015 έθεσε αυτό το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και γνωρίζουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει και άλλη μία εισήγηση το Μάιο του 2011 για το ζήτημα αυτό και θα ήθελα να προσθέσω ότι βιώνω, παρατηρώ μάλλον ότι υπάρχει ισχυρότατη ε, δέσμευση και από την προηγούμενη και την τωρινή και την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου. Ε, έχει αναδυθεί σε προτεραιότητα σε διάφορα θεσμικά όργανα αυτό το ζήτημα και για αυτούς τους λόγους είμαι πεπισμένη ότι τώρα από κοινού όλοι ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχει οριμάσει πια ο καιρός, ε, μπορούμε να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις πλέον. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να αναλάβουμε δράση για να καταπολεμήσουμε τη βία ε, που ασκείται κατά των γυναικών λόγω του φίλου τους. Ε, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία συζητούμε αυτό το θέμα της βίας ε, κατά των γυναικών και παρά την μεγάλη συνειδητοποίηση περί του ζητήματος αυτού ακόμη δεν έχουν αναλυθεί συγκεκριμένα μέτρα ε, που να έχουν ευοδοθεί και να έχουν ε, περιορίσει ή σταματήσει το φαινόμενο της βίας και γι' αυτό σας είπα ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε τώρα πρέπει να κινηθούμε, πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Η βία κατά των ε, γυναικών πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που πλήττει μόνο τα θύματα αυτών των βίαιων πράξεων. Μην ξεχνάτε ούτε για μία στιγμή ότι αυτή η βία πλήττει τις γυναίκες συλλογικά. Τις γυναίκες που απόσχουν από κάποιες επιλογές ζωής ε, διότι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο της βίας. Ε, δηλαδή η καθημερινή ζωή όλων των γυναικών περιορίζεται λόγω του φόβου ε, για τη βία, για τη σεξουαλική βία κτλ. Ε, πόσες ε, νεαρές κοπέλες επιλέγουν να μην κάνουν κάποια πράγματα διότι έχουν επίγνωση του κινδύνου που διατρέχουν. Αν παραδείγματο χάρη επιστρέψουν μετά το σινεμά στο σπίτι τους, μόνες τους. Περιορίζουμε δηλαδή τις επιλογές ζωής που κάνουμε διότι έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να αποφύγουν να περάσουμε στα σκοτεινά μέσα από ένα πάρκο παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ολόκληρη η ζωή μας ως ε, γυναίκες ε, διέρχεται, ε, περνάει με αυτή την επίγνωση, με αυτό το φόβο που διατρέχουμε μόνο και μόνο επειδή είμαστε γυναίκες. Είναι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα μέσα στην έκθεσή μου θα συμπεριλάβω διάφορες προτάσεις και θα ήθελα τώρα να επαναλάβω πως αυτή τη δουλειά θα την κάνουμε όλοι από κοινού στην Επιτροπή, ε, διότι γνωρίζω πόσο πολυάριθμα είναι τα μέλη της Επιτροπής ε, που έχουν πολλές γνώσεις στον τομέα αυτό και μπορούν ε, αποτελεσματικά να συμβάλλουν. Ε, στις εργασίες μας. Ε, έχουμε διεθνείς σε βάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ήδη αναφέρθηκα στις εργασίες και στις συμβάσεις και τα ψηφίσματα του Οργανισμών Ημένων Εθνών για αυτό το θέμα και θα ήθελα να τονίσω επίσης ε, τη νομική βάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ισότητα των δύο φύλων είναι μια θεμελιώδης αρχή της Ένωσης. Επίσης είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επίσης έχουν κέρια θέση μέσα στη συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα με την συνθήκη της Λισαβόνας αυξάνονται οι δυνατότητες μας για να κινηθούμε στον τομέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ε, μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε ποια μέτρα συγκεκριμένα πρέπει να αναλάβουμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πια τη νομική βάση, διότι έχουμε μία νομική βάση που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι έχουμε ευθύνη έχουμε, ε, ε υπάρχει ε, καθήκον ε, του κράτους να παρεμβαίνει όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κάποιων με πράξεις βίας ή σεξουαλικής βίας και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα της Στοκχόλμης Δηλαδή αναφέρομαι τώρα γενικότερα από ό,τι καταλάβατε στα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και βάσει του προγράμματος Στοκχόλμης ε, δυνάμεθα να αναλάβουμε κοινά μέτρα για να προστατεύσουμε τα θύματα πράξεων βίας. Ε, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τα όσα είπαμε για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, αυτό που ψηφίσαμε νωρίτερα σήμερα, σημαντικότατο εργαλείο για την προστασία των γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξεις από τη βία. Ο ορισμός τώρα της βίας λόγω φύλου ε, τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω ότι λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι πρόκειται για οποιαδήποτε πράξη βίας που οδηγεί ή, ή κατά πιθανότητα θα οδηγήσει σε ε, φυσικές, ε, ψυχολογικές ε, ή σωματικές ζημιές για τις γυναίκες ή όταν υπάρχει γενικότερη απειλή για τέτοιες βιοπράξεις ή όταν οδηγούν κάποιες πράξεις στέρηση της ελευθερίας είτε πρόκειται για πράξη. Ε, που λαμβάνουν χώρα σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό χώρο. Λοιπόν, η βία κατά των γυναικών συνιστά καταπίεση των γυναικών ως άτομα, αλλά και όπως σας είπα ε, νωρίτερα και ως σύνολο, ως κοινωνική ομάδα. Δεν χρειάζεται τώρα να κατονομάσω όλες τις μορφές ε, της βίας λόγω φύλου. Τα γνωρίζουμε όλοι. Ε, τα βιώνουμε όλοι στις χώρες όπου ζούμε και δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα. Όταν ανοίγουμε την εφημερίδα μας ε, βλέπουμε επιχαίως τίτλους ε, για δολοφονημένες γυναίκες για ενδοοικογενειακή βία, για εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστικούς γάμους και ούτω καθεξής. Όλες αυτές ε, οι μορφές ε, βίας ε, είναι οι διαφορετικές εκφάνσεις ενός ίδιου φαινομένου που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Εγώ κρίνω πως τίθεται ζήτημα αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών επίσης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. και θεωρώ ότι τα μέτρα κατά της βίας ε, δεν μπορούν να βασιστούν σε ένα μόνο παράγοντα. Ε, δεν θα αλλάξουμε με κάθε μέτρο έναν παράγοντα γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο, όλους τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν ε, στις βιοπράξεις. Ε, το θέμα της βίας κατά των γυναικών είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα διότι επισύρει κόστος ε, για την κοινωνία ε, λόγω των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργεί, κόστος για την περίθαλψη, για την απονομή δικαιοσύνης και μέσα στην έκθεση υπάρχει και μια εκτίμηση για το κόστος της βίας Ανά ώρα μέσα στα ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα κοστίζει η βία και ε, γι' αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό το στοιχείο. Είναι κοινωνικό πλέον το πρόβλημα εφόσον η βία επισύρει αυτό το επιπρόσθετο κόστος πάντως. Το βασικό είναι ότι τίθεται ζήτημα ισότητας. Κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να ζει ε, επαπειλούμενος μα, με αυτή τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του. Γυναίκες που ζουν σε τέτοιες ε, σχέσεις, η τραγωδία για κάθε παιδί που ε, βιώνει την ενδοοικογενειακή βία, ε, η ασφάλειά τους που τίθεται σε κίνδυνο, και βλέπουν τις βάναυσες αυτές πράξεις μέσα στην οικογένειά τους, οπότε ε, ε, ε, υπάρχει και πλήρης απώλεια της συναισθηματική σταθερότητας και ασφάλειας για αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά που βλέπουν αυτές τις πράξεις βίας ανάμεσα στους ενηλίκους, ανάμεσα στους γονείς τους. Κανένα παιδί θα έπρεπε να ζει υπό αυτές τις συνθήκες. Ε, τώρα για τις ε, οικογενειακές σχέσεις, συντροφικές σχέσεις, σας μίλησα για τα παιδιά. Και σε ορισμένε περιπτώσει ε, θεωρούμε ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Λέμε, α, ένα τσακωμό είναι ανάμεσα στο ζευγάρι. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό ιδιωτική υπόθεση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αγγίζει ολόκληρη την ε, κοινωνία και άρα συνιστά και ευθύνη ε, ολόκληρης της κοινωνίας ε, στις σχέσεις εγκύτας, συντροφικές σχέσεις, ε, η βία οδηγεί σε απομόνωση και η βία ή η απειλή βίας πλήττει τις γυναίκες και οι γυναίκες χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, νιώθουν άχρηστες, ανάξιες γιατί ε, εκτίθενται σε αυτήν την άποψη για τις ίδιες ε, ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και θεωρώ ότι θα πρέπει να αυτεπαγγέλτος να διώκεται μία τέτοια πράξη βίας διότι το θύμα ε, αυτής της ε, πράξης ε, δυσκολεύεται είτε να καταγγείλει ή το, την ίδια την αξιόπινη πράξη να εμείνει στην καταγγελία της. Συχνά δηλαδή αποσύρουν οι γυναίκες τις καταγγελίες τους διότι πλέον δεν, ε, πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να ζητήσουμε αυτεπαγγέλτος να διώκονται αυτές οι αξιόπινες πράξεις. Επίσης, να αναφερθώ σε μια άλλη κατάσταση που βιώνουν οι γυναίκες. Ε, Φερρυπίν ανάπηρες γυναίκες. Πόσο ελάχιστες δυνατότητες έχουν να ξεφύγουν από μια τέτοια σχέση. Σκεφτείτε, ε, έχουμε γυναίκες ε, τοξικομανείς, ε, γυναίκες άστιγες και ούτω καθεξής. Αυτοί η βία πλήττει όλες τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που είναι πιο εκτεθειμένες για άλλους λόγους και άρα δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση και χρειάζονται ακόμη περισσότερη βοήθεια από την κοινωνία για να τα βγάλουν πέρα. Σκέφτομαι αυτός που ζουν σε ιδρύματα ε, που δεν γνωρίζουν ε, ακριβώς το πώς έχει η κατάσταση για την ε, σεξουαλική βία και την σεξουαλική παρενόχληση είναι άλλο ένα θέμα που ε, συμπεριλαμβάνω στην έκθεσή μου γιατί η σεξουαλική βία πλήττει τις γυναίκες με λίγο καταστροφικό τρόπο και τίθεται ζήτημα εξουσίας, δηλαδή ε, τους αρνούνται στις γυναίκες το δικαίωμα για σεξουαλική ακαιρεότητα και για το δικαίωμα επιλογής Επίσης ακροτιαρισμός ε, των ε, γυναικείων γενετικών οργάνων και καταναγκαστική γάμη. Να άλλο ένα πρόβλημα που πλήττει τις γυναίκες και ελπίζω ότι και για αυτά τα ζητήματα θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ούτως ώστε να κάνουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις για να σταματήσουμε αυτά, αυτή τη βία. Ήδη ε, έχουμε ψηφίσει για το σχέδιο σχετικά με την εμπορία ανθρώπων το σχέδιο οδηγία για την εμπορία ανθρώπων και χαίρομαι που υπήρχε τόσο ισχυρή στήριξη από πλευρά της Επιτροπή. Ε, τέλο να σα πω ποια είναι η προσωπική μου τοποθέτηση για την εμπορία ανθρώπων και για την ε, πορνεία θα ήθελα να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για τις σχέσεις ανάμεσα στην νομοθεσία περί πορνείας στα διάφορα κράτη-μέλη και ε, το την ε, γενικότερη αντίληψη κοινή γνώμης για την εμπορία ανθρώπων. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα δύο, αλλά χρειάζονται πιο υπεριστατωμένες μελέτες για να το μπορέσουμε να το αποδείξουμε, οπότε καλό θα ήταν να επιζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Σας είπα και το ξαναλέω ότι πρέπει να διώκεται ε, αυτεπαγγέλτος οποιαδήποτε τέτοια αξιόπινη πράξη. Επίσης τα θύματα πρέπει να έχουν ε, το δικαίωμα να ζητήσουν νομική συνδρομή ε, γιατί δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται. Τη στιγμή της δίκης ο δράστης μπορεί να έχει δικηγόρο, ε, να έχει νομική συνδρομή και εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε το ότι τα θύματα της βίας επίσης ε, ε, θα ε, έχουν ε, το δικαίωμα αυτό, το δικαίωμα της νομικής συνδρομής. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν καλύτερη γνώση της κατάστασης. Μιλώ για όλες τις αρμόδιες αρχές, για την απονομή δικαιοσύνης, για την ιατρική περίθαλψη, η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ελπίζω να υπάρχουν εγχειρίδια, παραδείγματος χάρη για τις αστυνομικές δυνάμεις, ε, πώς ακριβώς ερευνούν ε, τέτοια εγκλήματα. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα κοινό εγχειρίδιο που πραγματικά να χρησιμοποιείται επί τόπου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είμαι πεπισμένη ότι με καλή ε, ε, συγγνώμη, καλή, σωστή εφαρμογή και χρήση του εγχειριδίου ε, δεν σημαίνει ότι προστατεύουμε μόνο τα δικαιώματα και κατοχυρώνουμε την προστασία του θύματος. Θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγχειρίδιο και για προληπτικούς λόγους, γιατί όσο περισσότερες γνώσεις, όσο περισσότερα ξέρουμε για αυτό το φαινόμενο, τόσο περισσότερο μπορούμε να επιτύχουμε σε επίπεδο πρόληψης. Ε, θα, θα, θα, κλείσω, θα σύντομα ε, γιατί θα συνεχιστεί και η συζήτηση. Ήθελα μόνο ε, να σας πω ότι μέσα στην έκθεσή μου προτείνω τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία ούτω ώστε να υπάρχουν ε, κέντρα προστασίας για τα θύματα Ε, πρέπει να, ε, για κάθε 10.000 κατοίκους να υπάρχει εφημερία ε, σε κάποιο τέτοιο κέντρο προστασίας θυμάτων. Αυτά τα κέντρα είναι μια βασική προϋπόθεση για κάποιον για να μπορέσει να φύγει από μια τέτοια βίαιη σχέση, για να έχει κάπου να πάει, για να προστατευτεί και αυτές οι εφημερίες ε, πρέπει να ε, στελεχώνονται με ε, κατάλληλα κατερτισμένο προσωπικό ανθρώπους που να μπορούν νομικός και αλέως να βοηθήσουν τα θύματα αυτά. Τέλος, τέλος, Α, το τηλέφωνο επίγουσα ανάγκη. Το συζητάμε αυτό το θέμα συχνά. Το είπαμε και για την εμπορία ανθρώπων. Λοιπόν, ε, ένα κοινό τηλέφωνο επίγουσας ε, ανάγκης για τα θύματα πράξεων ε, βίας λόγω φύλου. Κανά κάτι άλλο που μπορούμε να προτείνουμε. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν κατάλληλε οδηγίες προς το προσωπικό που θα απαντάει στο τηλέφωνο, που θα συζητά με τα θύματα. Επίσης, ενημέρωση μέσω διαδικτύου, το θύμα να μπορεί στο διαδίκτυο να δει ποιε δυνατότητε δυνατότητες υποστήριξης και αρρωγή υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Τέλος, οι δράστες, δράστες που διαπράττουν αυτά, αυτές τις αξιόπαινες πράξεις Είπα ε, προηγουμένως ότι πρόκειται για ε, έγκλημα, δίκημα, αξιόπινη πράξη και θα πρέπει να, ε, έτσι να αντιμετωπίζεται ενώπιον του δικαστηρίου. Θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους, ε, θεραπευτικές αγωγές ε, μέσω των συνεντεύξεων ε, για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά των δραστών, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να περάσουμε από δίκη, να δικαστεί αυτή η αξιόπινη πράξη πρώτα και μετά να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά του δράστη. Πολλοί έχουν εργαστεί για αυτό το θέμα και ε, το σημαντικό είναι να σπάσουμε τη σιωπή ε, για αυτή την βία. Αυτό που κάνουμε τώρα ε, τι είναι, συζητήσεις, διασκέψεις, με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για αυτό το φαινόμενο της βίας και σημαντικό είναι αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και δράσεις και επίσης Ε, επ' ευκαιρία της έκθεσης ε, συζητάμε το θέμα των γυναικών που είναι θύματα αυτής της βίας. Ε, ναι, τα πιο πολλοί άριθμα θύματα είναι οι γυναίκες, αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο θύματα της βίας οι γυναίκες, είναι πολλά περισσότερα. Πρέπει να δούμε και να δείξουμε σε αυτές τις γυναίκες που ζουν τη βία μέσα στη σχέση τους, μέσα στην οικογένειά τους, να δείξουμε σε αυτές τις γυναίκες ότι υπάρχει δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από αυτή την καταστροφική σχέση και πρέπει να δείξουμε ε, σε αυτές τις γυναίκες ε, ότι είναι δυνατές, ότι μπορούν μόνες τους να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή και για τις ίδιες και για τα παιδιά τους. Θέλω να τονίσω επίσης ότι όταν συζητούμε αυτό το θέμα της βίας λόγω φύλου, προσπαθούμε να τονίσουμε ότι γίνεται να ξεφύγουν αυτές οι γυναίκες, ότι γίνεται να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή για αυτές και για τις γυναίκες τους. Αυτό είναι σημαντικό να το καταδείξουμε στις γυναίκες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε όλοι μαζί από κοινού αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως σας είπα ήδη ανυπομονώ για τη μελλοντική συνεργασία που θα έχω και με τους συναδέλφους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Merci, Madame le rapporteur, de euh, cet exposé. Σας ευχαριστώ μας παρουσιάσατε ε, μας κάνατε μια πληρέστατη ε, παρουσίαση του ζητήματος και βλέπουμε πόσο αφοσιωμένοι είστε σε αυτόν τον αγώνα. Ε, η κυρία Γκαρσία Περές και η κυρία Μπιλμπάου ακολουθούν. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνάδελφος η κυρία Εστρέλα είναι σκιώδης συγγήτρια της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παραστεί. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, πρέπει να παρίσταται σε άλλη συζήτηση και κάποια θέματα θα ήθελα να διαβιβάσω σε σχέση με τοποθετήσεις της. Πρώτα απ' όλα φυσικά να συγχαρώ για το έργο που έχει υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό πιστεύω, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και με την πεποίθηση που διαβιβάζεται το έργο αυτό και διαχέεται από την Επιτροπή στην οποία εργαζόμαστε αληθεύει ότι αρκετές ευκαιρίες είχαμε που μπορούσαμε να θέσουμε την ανάγκη και να την εκφράσουμε να εμπλακούμε περισσότερο και να εργαστούμε περισσότερο σε όλα τα θέματα που αφορούν ε, την καταπολέμηση της βίας του φύλου, της βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της σε μια άνηση κοινωνία. Αυτή είναι η πεμπτουσία. Επ' αυτού πρέπει να εργαστούμε. Οι γυναίκες που είναι θύματα της βίας, α, είναι θύματα της βίας για το γεγονός ότι είναι γυναίκες. Γιατί οι άντρες πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι πάνω από τις γυναίκες και η βία του φίλου, εις βάρος των γυναικών πρέπει να αντιμετωπίζεται εγκάρσια, οριζόντια. Υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν τα θέματα. Όπως όμως το αναφέρει και η έκθεση, τη νομική βάση την έχουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό μέσα σε αυτή την έκθεση το ότι έχουμε μια νομική βάση και έτσι μπορούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε στην ε, μάχη της καταπολέμησης της βίας του φύλου, βίας εις βάρος των γυναικών, με διάφορα μέσα. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια οδηγία κατά της ε, βίας του φύλου, κατά της βίας των γυναικών, είναι διαφορετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου αυτή η νομοθεσία όπως στην Ισπανία, στη χώρα μου, είναι σαφέστατη, κάθετη. Υπάρχει ε, νομοθέτημα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Χαρακτηρίζεται έγκλημα και υπάρχουν πολλά μέσα για να καταπολεμηθεί. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες όπου αυτή η δουλειά δεν ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μέσα που θα είναι κοινά κοινά εργαλεία. Χρειαζόμαστε κοινά στοιχεία επίσης που είναι πολύ σημαντικά, θεμελιώδους σημασία. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στι οικονομικέ επιπτώσει που έχει η βία ει βάρο των γυναικών και είναι θεμελιώδες να μπορέσουμε να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία και στοιχεία ομοιογενή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να έχουμε μια αξιολόγηση σφαιρική και συνολική όσον αφορά αυτό το θέμα είναι σωστή επίση και η αναφορά που γίνεται στην ανάγκη του να δρομολογηθεί ένα παρατηρητήριο κατά τη βία ει βάρο των γυναικών στου κόλπου του Ιδρύματο για τις γυναίκες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοβουλία που αναλήφθηκε και προάχθηκε από την Ισπανική Προεδρία. Πρέπει να πάρει σάρκα και οστά αυτό το μέσο. Μπορεί να εξυπηρετήσει όλου μα για να δρομολογηθούν διαφορετικέ πρωτοβουλίε, ιδιαίτερα σε αυτή την ανάλυση, μελέτε, στοιχεία που θα συλλέγονται και θα αναφέρονται σε αυτό το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Θα είμαι σύντομη επειδή έχουν πολλοί ζητήσει τον λόγο, πολλές έχουν ζητήσει τον λόγο. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την διαθεσιμότητα και την προθυμία και θα πρέπει να εργαστούμε σε κάποιες πτυχές για να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο σε όλα αυτά τα θέματα σφαιρικά. Πιστεύω ότι η ψηφοφορία σε σχέση και η ομόφωνη τοποθέτηση και για την ε, εντολή προστασία και για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών δείχνει ότι από κοινού πρέπει να εργαστούμε οι γυναίκες να δώσουμε το παράδειγμα να προχωρήσουμε σε τόσο σημαντικά θέματα για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Merci, Madame Garcia Perez. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκαρθία Πέρεθ και η κυρία Βιμπά θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον τρόπο που ε, παρουσιάστηκε και στην η έκθεση. Εγώ σε σχέση με αυτήν την έκθεση θα ήθελα να πω ότι όταν κάνουμε λόγο για την εστίαση, την επικέντρωση, τη σφαιρική, εκείνο που μου λείπει είναι ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και κάποιες άλλες πτυχές, όχι μόνο αυτές που συσχετίζονται με τη βία. Και αυτό γιατί, διότι Ίσως επίσης επειδή όπως ανέφερε η κυρία Γκαθία πιο πριν αν υφιστάμεθα βία οι γυναίκες από τους άνδρες είναι επειδή είναι άνηση η κοινωνία. Η σφαιρική αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έπρεπε να μας κάνει να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι ανισότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές που άμα συνειδητά τις αντιμετωπίσουμε μας οδηγούν σε αυτή την έκρηξη βίας, σε αυτές τις καταστάσεις έκδηλης βίας. Και το 2005 στην αυτόνομη περιοχή των Βάσκων υιοθετήσαμε ένα νομοθέτημα σφαιρικό, συνολικό και με αυτή την επικέντρωση νόμος ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφέρεται αυτό το νομοθέτημα και υπάρχει ένα εδάφιο όπου αναφέρεται γιατί υπάρχει ανισότητα και αναφέρονται τα εργαλεία και τα μέσα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε αυτή τη βία. Η επικέντρωση στο κείμενο του ψηφίσματος είναι ότι θα πρέπει αυτό να λάβουμε υπόψη και γι' αυτό κάπως ε, έχω, ε, διαφέρουμε σε σχέση με το κείμενο του ψηφίσματος. Από εκείνο το σημείο λοιπόν, οι ίδιες οι πρωτοβουλίες και για το ίδιο το κείμενο του ψηφίσματος θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια πιστεύω για να αναλύσουμε και να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν είτε σε άλλες χώρες είτε σε άλλες περιοχές και περιφέρειες. Διότι πραγματικά υπάρχουν παρατηρητήρια καταπολέψεις της βίας που λειτουργούν. Υπάρχουν αριθμοί κλήσεις τηλεφωνικοί που λειτουργούν. Υπάρχουν πρωτόκολλα δράσης ε, νομοθετικά, δικαστικά, αστυνομικά υγειονομικά που στοχεύουν πρώτα απ' όλα σε πρώτο, κατά πρώτο λόγο να αναπτύσσουν σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς δράσεις ώστε να συντονίζονται και όταν υπάρχει περίπτωση βίας να ενισχύονται και από την κατάρτιση και ε, παιδεία, εκπαίδευση του προσωπικού, είτε του αστυνομικού, είτε του υγειονομικού προσωπικού, του δικαστικού. Έτσι, σε σχέση με την παρατήρηση που έκανε η ίδια η πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προσπαθώντας να δώσουμε συγκεκριμένη μορφή σε αυτά, διότι υπάρχουν εμπειρίες. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις ε, δρατώμενοι της γνώσης που υπάρχει και να δούμε όλες ή όλοι μας αν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι καινοτόμο. Είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την πορεία να συμπεριλάβουμε τους άντρες. Δεν θα πετύχουμε την ισότητα αν δεν εργαστούμε από κοινού γυναίκες και άντρες και θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού ε, οι γυναίκες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι μια προσέγγιση, μια επικέντρωση που πρέπει να προχωρήσουμε. Στην πορεία αυτή, στη διαδρομή, να μας βοηθήσουν οι άνδρες και να μας συνοδεύσουν, γιατί θα είναι καλό και για αυτούς. Ένα άλλο θέμα, όταν κάνουμε λόγο για τις καταγγελίες, για τις ε, τράπεζες δεδομένων και τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται, συμφωνώ, πρέπει να έχουμε στατιστικά στοιχεία εξειδικευμένα, να γνωρίζουμε το θέμα για να το αντιμετωπίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Όταν κάνουμε λόγο για δολοφονημένες γυναίκες, θα ήθελα να συμπεριλάβουμε επίσης τα στοιχεία των παιδιών που ε, αγοριών και κοριτσιών που είναι και αυτά θύματα της ε, οικογενειακής βίας και πολλές φορές δολοφονούνται παιδιά, κορίτσια, γη που δολοφονούνται από κοινού με τις μητέρες τους. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτή τη διάσταση ακριβώς των παιδιών θυμάτων και να δώσουμε μια προοπτική επίσης πιο σύγχρονη του 21ου αιώνα σε αυτά διότι βλέπουμε και ζούμε ότι έχουμε νέες μορφές ζευγαριών τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια που επαναλαμβάνουν τις ίδιες μορφές βίας, τις ίδιες περιπτώσεις βίας σαν αυτές που υφίστανται οι γυναίκες. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πραγματικότητες σε αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε υπόψη μας. Και επίσης να πω κάτι άλλο, ότι υπάρχει, υπάρχουν επίσης τοπικά δίκτυα που λειτουργούν μέσω ε, δικτύων περιοίκων και ε, συνοικιών. Στην ε, περιοχή των Βάσκων έχουμε με, μέσω δικτύων δήμων και κοινοτήτων στη χώρα των Βάσκων προσπαθούμε να εκπονήσουμε τέτοια στοιχεία συγκεκριμένα και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι συμφωνώ με όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν σε σχέση με τη ζημιά που, προκαλούν, που προκαλείται από τις διάφορες μορφές βίας. Το δικό μας προτέρημα πρέπει ως Κοινοβούλιο να είναι να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερες συγκλήσεις και μεγαλύτερη, ε, ας έτσι, ε, μεγαλύτερο συντονισμό. Πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες αρρωγής και ε, συνδρομής. Αλλά πρέπει επίσης και ένα άλλο θέμα να δούμε. Τις νομικές υπηρεσίες ή δικαστικές αστυνομικές υπηρεσίες που πρέπει να ε, εξετάζουν αυτές τις καταγγελίες και να δίνουν συνέχεια. Αλλά υπάρχουν ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα που ζούμε καθημερινά και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αποσύρονται τόσες καταγγελίες από τις γυναίκες ενώ έχουν διατύπωθεί αρχικά. Όχι μόνο επειδή, δεν υπάρχουν, ε, ε, επειδή οι κοινωνικές υπηρεσίες πολλές φορές όπου παρουσιάζονται αυτές οι καταγγελίες μετά οι γυναίκες τις αποσύρουν. Τι συμβαίνει. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και σαν ένα πρόβλημα εξάρτησης. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Για αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις που γνωρίζω, οι γυναίκες με εντάλματα προστασίας αποσύρουν πολλές φορές καταγγελίες ή αφήνουν περιθώριο, ας το πω έτσι, στον ε, ε, θήτη αφήνουν ε, το πεδίο ελεύθερο στο θήτη. Πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω για την περιεκτική έκθεση που συνέταξε η, η συγγήτρια και πρέπει να συνεργαστούμε για να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο στην ευρωπαϊκή κοινωνία την ευκαιρία να μην είναι τα, οι γυναίκες θύματα και να μην αποτελούν αντικείμενο ε, έκδηλης βίας. Ευχαριστώ. Merci, Madame Bilbao. Ε, ευχαριστούμε, κυρία Μπιλμπάου. Η κυρία Τσέσκοβα τώρα. Děkuji ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, να την ευχαριστήσω και παρότι ε, είμαι σε αυτή την Επιτροπή για αρκετό διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα λίγα θέματα, πρέπει να ομολογήσω, όχι το μόνο, αλλά ένα από τα λίγα θέματα και αντικείμενα που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά μου. Δεν θέλω να υποτιμήσω το έργο άλλων εισηγητριών και εισηγητών, αλλά αυτό βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά αυτού που θα έπρεπε να αναπτύσσει ως έργο η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θεωρώ και πιστεύω ότι αν οι γυναίκες χρειάζονται προστασία, είναι η προστασία κατά της βίας αυτή η προστασία που χρειάζονται. Σε προηγούμενες δηλώσεις μου αυτό που είχα αναφέρει ήταν είχα αναφερθεί σε γυναίκες μόνες που ανατρέφουν τα παιδιά τους και ε, αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και θέματα ε, παινίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα που εμείς σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα έπρεπε να αναπτύξουμε και να αναλύσουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο του έργου μας. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έχει πραγματικά σταθε, αξιόπιστη και σταθερή νομική βάση. Οι ιδέες που ε, συμπεριλαμβάνονται είναι σαφείς, περιεκτικές και εκφράζονται με έναν τρόπο θα έλεγα πραγματικά ε, πιστικό. Παρόλα αυτά θα ήθελα από την άλλη πλευρά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια. Σχόλια που βασίζονται σε αυτά τα οποία ακούσαμε στις ε, ενακτήριες ε, αρχικές παρατηρήσεις της εισηγήτριας και μετά από παρατηρήσεις που ακούστηκαν στη συζήτηση. Πρώτα, όταν έρχεται η ώρα της προστασίας της αναπαραγωγικής υγείας όπως ε, καθορίζεται από τον, τον, τον, ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είμαι υπέρ βέβαια όσον αφορά τέτοια δράση. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει και να εντάσσεται σε όλες τις εκθέσεις τέτοιου τύπου και χαρακτήρα. Είναι κάτι το οποίο αναφέρατε κυρία εισηγήτρια στον λόγο σας και είναι κάτι το οποίο πάντα θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και να υποστηρίζουμε. Αν οι γυναίκες θέλουμε να είναι ελεύθερες, τότε θα πρέπει να είναι ελεύθερες πάνω απ' όλα για να αποφασίζουν για θέματα της υγείας τους οι ίδιες Υπάρχουν τώρα κάποια ε, σημεία τα οποία επέλεξα σε σχέση με την έκθεση. Λυπούμε πολύ που δεν ήμουν σε θέση να παραστώ στην ακρόαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Γνωρίζω ότι διεξήχθη μία ακρόαση την Τετάρτη. Ήταν ιδιαίτερα φορτωμένη όμως αυτή η προηγούμενη εβδομάδα της περίοδου συνόδου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου και δεν μπόρεσα να παραστώ. Παρ' όλα αυτά όμως, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στην παράγραφο 6, αν δούμε το κείμενο, ελπίζω ότι θα μπορούσα να πείσω την ομάδα μας να τροποποιήσει τη διατύπωση σε σχέση με, αυτό το, με αυτή την παράγραφο. Και αυτό επειδή δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε τόσο περιορισμένοι όσον αφορά ένα τόσο αυστηρό όριο όσον αφορά τις δομές και η παράγραφος 7 που αφορά την πορνεία. Το αναφέρατε αυτό εξάλλου και στην παρέμβασή σας και συζητήθηκε και στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων κιόλας αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα της πορνείας. Εγώ προσωπικά πιστεύω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι θα έπρεπε ότι καλό είναι να απαγορευτεί η, άσκηση της πορνείας μάλιστα νομικά με νομοθέτημα αλλά αυτό θα έπρεπε απλά να μας κάνει να δούμε ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλαίσιο απαγορευτικό, αυτό θα οδηγούσε στο, στις γυναίκες να οδηγούνται στο να κρύβονται μετά και τα θύματα θα ήταν ας το πω έτσι άφαντα και αόρατα και θα υπέφεραν ακόμα περισσότερο εφόσον θα κρυβόντουσαν. Γι' αυτό τόνισα ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της παραγράφου 7 στην έκθεσή σας και είμαι ευγνώμων σε εσά για αυτή την έκθεση. Σίγουρα όμως από την άλλη πλευρά ανεκδοτολογικά θα ήθελα να πω ότι κάνατε λόγο για την βία, άσκηση βίας μέσα στο, στις σχέσεις ενός ζευγαριού. Όμως αυτή η έννοια με την οποία δεν, ε, ε, δεν είχα εξοικειωθεί παρότι βέβαια ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ο σύζυγός μου με κατηγορεί ε, στο σπίτι μας. Δεν θα ήθελα λοιπόν αυτό να είναι μια ε, καταδικαστέα πράξη, διότι το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν ο σύζυγός μου να με προσάξει στα δικαστήρια. Λέει ότι εγώ τον υποχρεώνω, λέει, να κάνει διάφορα πράγματα, όπως αυτά τα οποία εσείς περιγράφατε ως βία εις βάρος των γυναικών. Παραπονείται εκείνος, ο σύζυγος τώρα. Πέρα από αυτό το ανέκδοτο, θα ήθελα σοβαρά τώρα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο το οποίο αναπτύσσεται εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσέσκοβα. Η κυρία Πλάμ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι εκτιμώ ιδιαίτερα την προσέγγιση αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρουμανία εμείς ξεκινήσαμε μία εκστρατεία με θέμα την ε, ενδοοικογενειακή βία η οποία αφορά όλους. Διότι το φαινόμενο αυτό επεκτείνεται όλο και περισσότερο και επεκτείνεται λόγω ε, των κοινωνικών ανισοτήτων. Βεβαίως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλε τα μάλα στην επέκταση αυτού του φαινομένου. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι ανεξάρτητα από το τι σημαίνει μέσα στην οικογένεια, όταν χάνει κανείς τη δουλειά του, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν πλέον τα προστοζήν. Γι' αυτό εκφράζουν μια επιθετικότητα για μένα λοιπόν βία σημαίνει άσκηση. Βία σημαίνει άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Και αυτό είναι μια επίθεση και στο μέλλον με την έννοια ότι μέσα σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγάρι όπου υπάρχουν μόνιμα καυγάδες Τελικά τα παιδιά είναι εκείνα που υποφέρουν περισσότερο. Και τα παιδιά είναι εκείνα που ε, πλήττονται και οι επιπτώσει θα φανούν στο μέλλον. Η βία λοιπόν είναι... έχει αποτελέσματα, έχει συνεπακόλουθα μάλλον και κατά τη δική μου άποψη η βία είναι άρρηκτα συνδεμένη με την φτώχεια, αυτό το ανέφερα και στην έκθεση που συζητήσαμε προηγουμένως. Ένας άλλος λόγος γιατί ασκείται βία είναι κατά την άποψή μου η έλλειψη παιδείας. το χάρη στη Ρουμανία έχουμε στατιστικά δεδομένα ε, για τη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά ε, τεκμηριώνουν αυτό που σας προηγουμένως ότι επεκτείνεται το φαινόμενο υπάρχουν πολλά θύματα που δεν έχουν το θάρρος να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν την άσκηση βίας που δέχτηκαν. Δεν έχουν το θάρρος να πούν στις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς συνέβη. Πιστεύω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα χρηματοδότησης για εξτρατείες πρόληψης και για την ε, δημιουργία ε, υπηρεσιών, για ε, παροχή υπηρεσιών, ε, παροχή συμβουλών για τα παιδιά. Υπάρχουν ε, καταφύγια όπου μπορούν να καταφύγουν τόσο οι μητέρες όσο και τα παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ ένα τέτοιο καταβλισμό στη χώρα μου. Όπως σας είπα λοιπόν, τα κράτη-μέλη οφείλουν να χρηματοδοτήσουν τις ΜΚΟ που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου της άσκησης βίας εις βάρος των γυναικών που όπως σας είπα το φαινόμενο διγκώνεται όλο και περισσότερο. Θέλω να σας ε, συγχαρώ για, την, ε, για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε το θέμα. Η ε, συνεισφορά σας είναι καθοριστική σημασίας. Και όσον αφορά Σα συγχαίρω επίση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το πώ πρέπει να ε, τύχει διαχείριση το φαινόμενο αυτό στην Ευρώπη. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θα αναλώσω πολύ, χρειάζεται να αναλώσω πολύ από τον χρόνο σας. Από πλευρά σας Βένσον, και εγώ η ίδια εδώ και χρόνια εργαζόμαστε και γνωριζόμαστε και ξέρω πόσα πόσες μάχες, πόσους αγώνες έχει δώσει κατά της βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών. Ξέρω το έργο που έχει επιτελέσει και πόσο θετικό είναι και θέλω να τη συγχαρώ για την έκθεση αυτή. Τώρα, πρόσφατα, συχνά κάναμε λόγο για τα θέματα βίας εις βάρος των γυναικών αρκετά κράτη-μέλη επενδύουν στο να βοηθηθούν τα θύματα και όσον αφορά την αστυνομία και την νομοθεσία καταβάλουν προσπάθειες να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ακούσω όμως περισσότερα για την πρόληψη. Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Ακόμα και ίσως και σε αυτή την έκθεση να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Διότι στις 20 παραγράφους μόνο μία αναφέρεται στην πρόληψη. Φυσικά από πλευρά μου είμαι ιατρός και αυτό τι σημαίνει. Αυτό ίσως σημαίνει ότι η πρόληψη είναι ακριβώς μια δεύτερη φύση όσον αφορά το άτομό μου. Αυτό προσυδειάζει στους γιατρούς. Όμως θεωρούμε και πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία επειδή και κοστίζει λιγότερο, είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή η πρόληψη. Αυτό που θα έπρεπε να σκεφτούμε περισσότερο να πετύχουμε είναι να σκεφτούμε τα οικονομικά ωφέλη του να κάνουμε κάτι παραπάνω για να προκαταλάβουμε, να προλάβουμε την έκρηξη βίας εις βάρος των γυναικών. Φυσικά αυτό θα σημαίνει λιγότερες ανθρώπινες ζωές που θα θυσιάζονται και θα καταστρέφονται πέρα από τα άλλα ωφέλη. Πρόσφατα όμως δεν έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό αρκετά πράγματα γιατί υπάρχει αυτή η βία εις βάρος των γυναικών και υπό ποιου όρους εκφράζεται και εκδηλώνεται και πώς. Η κυρία Πλούμπ αυτό που έκανε είναι ανέφερε τη φτώχεια, το ενόπνευμα, το αλκοόλ, τα ε, ε, ναρκωτικά και την Ζήλια που είναι οι τέσσερις κύριοι λόγοι, οι τέσσερις κυριότεροι λόγοι που αποτελούν μέρος ε, του, των εξηγήσεων και των λόγων αυτών των πράξεων βίας ε, που παρατηρούνται εις βάρος των γυναικών. Γι' αυτό πιστεύω ότι ε, έλλειψη σεβασμού για την αξιοπρέπεια των γυναικών και αυτό αποτελεί μέρος αυτής της εξίσωσης ή απουσία σεβασμού της αξιοπρέπειας των παιδιών εξίσου. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις χαρακτηριστικά που οδηγούν στην βία εις βάρος των γυναικών να είναι πιο έντονη και πιο πιθανή. Και όπως ε, ε, υιοθετούμε στρατηγικές και εκστρατείες ε, κατά της βίας εις βάρος των γυναικών πρέπει να δράσουμε και προληπτικά. Έχει αποδειχθεί ότι παιδιά που ανατρέφονται και μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βίας πιθανότατα αυτά τα ίδια τα παιδιά θα γίνουν βίαιοι ενήλικες ε, και θα ασκούν βία ως ενήλικες. Είναι λοιπόν τρομερό το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά ώστε αυτά τα ίδια τα παιδιά να μην είναι βία έναντι των ε, εταίρων και συντρόφων τους ε, όταν είναι πλέον ενήλικοι. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να επιμείνω κι εγώ για κάποια ζητήματα που με ενδιαφέρουν όλος ιδιαιτέρως σε αυτόν τον αγώνα ε, κατά της βίας και για τη γενικότερη κινητοποίησή μας. Πρώτον, ο στόχος να σπάσουμε τη σιωπή, είπαμε. Τελικά δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη βία παρά μόνο όταν γνωρίζουμε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό, αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε τίποτα, καμία πτυχή. Να σπάσουμε τη σιωπή, ούτως ώστε όλα τα θύματα βίας να μπορέσουν να εκφραστούν. Αν το πετύχουμε αυτό, θα συνειδητοποιήσουμε ότι η βία υπάρχει σε όλες τις ε, κοινωνικές ε, τάξεις. Και είναι πολύ ε, δύσκολο να παρεύουμε ακριβώς λόγω της ευρύτας εμβέλειας του προβλήματος. Υπάρχουν ε, περιβάλλοντα, τάξεις όπου είναι πολύ προφανέστερη η βία σε σχέση με ε, άλλες και δεν είναι εύκολο να οριοθετήσουμε το πρόβλημα. Θέλουμε να φτάσουμε στην καρδιά, στη ρίζα του προβλήματος. Θα πρέπει να σπάσουμε τη ε, σιωπή και να ε, παρισφρήσουμε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, παρότι για κάποιους ε, θα είναι δύσκολο να παραδεχτούν ότι είναι βίαιοι. Δεύτερον, αλλά το προανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι μεταξύ των οποίων κυρία Ζαμπόσκα, πρέπει να είμαστε σε ε, γρήγορωση σχετικά με τις επιπτώσεις της βίας ανάμεσα στους γονείς επί των παιδιών. Γιατί όχι μόνο υπάρχει μια ψυχολογική καταστροφή, μια βαθιά ψυχολογική ανασφάλεια στα παιδιά των οποίων ε, οι γονείς ζουν αυτό το φαινόμενο, αλλά συχνά υπάρχει και επανάληψη αυτών των πράξεων διαγενειακή. Και πάλι εδώ, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δράσεις που θα μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε ε, τη, την κατάσταση. Ε, και κυρίως για να προλάβουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, το σωστά θέσατε το ζήτημα του κόστους ε, της δράσης αλλά και η πρόληψη έχει θεμελιώδη σημασία και νομίζω ότι έχουμε μεγάλο περιθώριο για να ενισχύσουμε τις προληπτικές δράσεις μας. Τρίτον, το τρίτο σημείο που θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή όλων είναι το ότι σε μια επιτροπή όπως η δική μας είναι λίγο δύσκολο να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα αλλά θα πρέπει ε, να ε, το συζητήσουμε, να συζητήσουμε το θέμα της ε, κοινή προσέγγισης, ενοποιημένης προσέγγισης. Δηλαδή να σκεφτόμαστε με διαυγή τρόπο γιατί να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι η βία δεν πλήττει μόνο τις γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες που δρούν βία κατά των ανδρών και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε άσπρα ή μαύρα τα... Ε, ζητώ συγγνώμη, έτσι μπορεί να δυσαρεστώ, να θορυβώ κάποιους με αυτά που λέω, αλλά ήρθε η στιγμή να το πούμε ε, σε διαζύγια παραδείγματος χάρη ε, ενδέχεται να υποστούν βία και οι άντρες όπως και οι γυναίκες. γνωρίζω ε, ε, περιπτώσεις ψυχολογικής λαιλασίας αν θέλετε κατά των ε, αντρών. Ε, ε, και νομίζω είναι, θα είναι προς τιμή μας ε, να έχουμε μια συνολική θεώρηση όλων των εκφάνσεων της βίας. Και δεν είναι μόνο προς τιμή μας, είναι αυτό που θα εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί ε, στην καταπολέμηση της βίας, ε, πρέπει να είμαστε διαυγείς, να είμαστε ανοιχτή και ε, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη για αυτό το ζήτημα. Τέλος, στα συγκεκριμένα μέτρα που πολύ ορθά ε, εκθέσατε, κυρίως αυτό που μας είπατε για τα κέντρα υποδοχής των θυμάτων, αλλά πέρα από τα κέντρα υποδοχής χρειαζόμαστε και μέσα για να λειτουργούν σωστά εύρυθμα αυτά τα κέντρα ε, σε κάποια κράτη σήμερα. Ε, μπορεί να υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής αλλά αν δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα για να λειτουργήσουν σε τι ωφελούν αν ε, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές ε, στρατηγικές θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους και να συνοδεύσουμε τη βούλησή μας από μέτρα. Η κυρία Πίκ τώρα θα πάρει το λόγο εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκω εδώ ε, μαζί με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη ε, και ήδη αναφερόμεθα στην εκπρίσωπο κυρία Ρέντινγκ η οποία έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση της ενδοικογενειακής βίας. Η δική μου λοιπόν η Γενική Διεύθυνση με αυτή τη δικαιοσύνη συνεργαζόμαστε στενά και από τον Ιανουάριο θα είμαστε και όλοι σε μια Γενική Διεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο της έκθεσης, ε, για την εισαγωγή της, να ευχαριστήσω ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τα σχόλιά τους και στηρίζω ανεπιφύλακτα την άποψη της ηγητρίας ότι η βία ε, που έχει σχέση με το φίλο ε, δεν σημαίνει, δεν είναι κάτι που πρέπει να γνωρείτε. Έχει ε, προεκτάσεις και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια δημόσια απάντηση. Ε, την περασμένη εβδομάδα πολλοί από εσά ήταν εδώ, είχαμε μια συνδιάσκεψη, ένα συνέδριο και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια μελέτη ε, που μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάστηκε από την Επιτροπή και είχε ως αντικείμενο το, την ανάγκη να εναρμονιστούν ε, οι εθνικοί κανόνες. Η δική μου η διεύθυνση παρουσίασε τα μέτρα που ελήφθησαν ε, σε όλα τα κράτη-μέλη για την πίεση βάρο των γυναικών. Πολλά λοιπόν παραδείγματα τα οποία σας παρουσιάστηκαν και γι' αυτό ε, συστήνω να ξαναδείτε το υλικό αυτό και είμαι σίγουρη ότι και η συγκήτρια θα το λάβει υπόψη της πριν ολοκληρώσει την έκθεσή της. Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και το είπαμε ήδη και στο Πεκίνο πριν από 15 χρόνια στη συνδιάσκεψη των Εθνών, ε, η βία εις βάρος των γυναικών σημαίνει ότι αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη στρατηγική, βεβαίως και συγκεκριμένα μέτρα. Η Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ την περασμένη εβδομάδα ε, στην αρκετή ομιλία της ε, ε, σε, αυτή την συνδιάσκεψη αναφέρθηκε σε μέτρα τα οποία θα υποβληθούν το Μάιο του επόμενου έτους. Αναφέρθηκε και σε μέτρα για την ισότητα των δύο φύλων και τις ενέργειες που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Δάφνη. Όπως ξέρετε η βία ε, που χαρακτηρίζεται από τη διάσταση του φύλου αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες μας και σχετίζεται και με άλλες προτεραιότητες. Όπως είπα προηγουμένως η πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρχει οικονομική ανεξαρτησία. Δίδοντας γυναίκες στην οικονομική ανεξαρτησία παρότι δεν σημαίνει ότι αυτές δεν θα δεσμευτούν σε ενδοοικογενειακή βία ε, σημαίνει ότι αν θέλουν μπορούν να ξεφύγουν. Βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλά αίτια, ε, πολλά ε, στοιχεία της ε, βίας που χαρακτηρίζεται από τη διάσταση του φύλου που δείχνουν ότι μπορεί να βρεθεί μια σωστή απάντηση. Η βία αυτή αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλες τις ομάδες της κοινωνίας μας και γνωρίζουμε επίσης ότι και κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Οι γυναίκες Ρωμά, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ευάλωτες. άκουσα ε, πριν από μερικές ημέρες για τις εμπειρίες που αντιμετωπίζουν και γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικέ ε, μορφές ε, καταβλισμών που να είναι προσαρμοσμένες σε αυτές γιατί αυτές δεν μένουν σε ένα και μόνο μέρος. Επίσης χρειαζόμαστε στις πολιτικές μας που ε, χαράσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ειδικές ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βίας με τη διάσταση του φύλου. Πρέπει βέβαια να έχουμε και μια ευρύτερη προσέγγιση και χαιρετίζουμε την πρόοδο στο Συμβούλιο της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της ε, σύμβασης. Ελπίζουμε να ε, λάβει μια συγκεκριμένη μορφή η εργασία αυτή σε συνεργασία με τα κρατημέλη για να καταστεί δυνατόν να εφαρμοστεί η σύμβαση. Γνωρίζω ότι παράλληλα θα υπάρχουν και πολλές συζητήσεις για το αντικείμενο. Και ένα από αυτά που έφτιαξε το Προεδρείο είναι ότι μιλάμε συνέχεια για την ενδοοικογενειακή βία που σημαίνει ότι η βία μπορεί να είναι είτε θηλυκή είτε ανδρική. Επάνω μιλάμε για τη βία που χαρακτηρίζεται από το διάσταση του φύλου και στο Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στα κράτη-μέλη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βία και τα αίτια της. Αλλά γνωρίζω επίση ότι μερικέ φορέ η γλώσσα είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση αναγνωρίζει και αυτό αναφέρεται ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπό την Ισπανική Προεδρία. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινά μέτρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδοοικονομική βία. Αυτό βέβαια γίνεται πολύ πιο εύκολα ε, από λέγεται πιο εύκολα από το να επιτευχθεί. Πάντως ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, συγκεκριμένες πολιτικές και στο μέλλον στο Βιλνιούς ε, το ειδικό αυτό Ινστιτούτο θα συνεχίσει να εξετάζει την εφαρμογή όλων των στοιχείων, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να γνωρίζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι ε, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να μάθουμε, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα και έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε το τι πρέπει κατά κύριο λόγο να μετρηθεί. Ελπίζω και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί η συγγήτρια στην έκθεσή της. Ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία με εσά κατά τους επόμενους μήνες και χαίρο για άλλη μια φορά ε, την συγγήτρια και την Επιτροπή για το θέμα το οποίο μας παρουσίασε. Σας ευχαριστούμε κύριε Βίκα. Τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια μας, την κυρία Σφένσεν, για να κάνει τα καταληκτικά της ε, σχόλια. Ένα θερμό ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω σε όλους τους συναδέλφους και φυσικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Όπως είπα στις αρχικές παρατηρήσεις μου, το θέμα της βίας λόγω φύλου ε, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων ε, και ενημερώθηκα πραγματικά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι δηλαδή δεν, χρειάζεται, ε, δεν χρειάζονται μεμονωμένα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα μια σειρά μέτρων πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και όπως είπαν οι συνάδελφοι, η βία αυτή οφείλεται στο ότι υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης στην κοινωνία μας και αυτό είναι ένα ε, θέμα που πρέπει φυσικά να απασχολήσει κατά προτεραιότητα την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας. Επίσης, ε, ε, είπαν οι συνάδελφοι ότι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα βίας, ότι είναι θέμα εξουσίας, θέμα ελέγχου ότι παρατηρείται το φαινόμενο σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Κάποιοι παράγοντες μπορούν δεν να έχουν καταλητική σημασία, όπως είδαμε, η φτώχεια, το αλκοόλ, η ανεργία και ούτω καθεξής. Μπορεί να, έχουν, να είναι καταλητικοί αυτοί οι παράγοντες, αλλά μην ξεχνάμε ότι η βία παρατηρείται σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις τάξεις, αλλά υπάρχουν όντως κάποιοι παράγοντες ε, που μπορούν να δράσουν καταλητικά και να οδηγήσουν σε αυτά τα φαινόμενα βίας. Επίσης μιλήσαμε για βέλτιστες πρακτικές και για ένα καλύτερο συντονισμό αυτών των βελτίστων πρακτικών και εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε ε, κάποια κοινή λύση. Επίσης μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ισότητας ε, των Δύο Φύλων. Φυσικά μπορεί να συμβάλλει και πρέπει να συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είναι βασικός φορέας στο όλο εγχείρημα. Ε, και ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα εκπονήσει μελέτη συγκεκριμένα όπου ε, θα ερωτηθούν γυναίκες από όλα τα κράτη-μέλη και για τα προσωπικά τους βιώματα σχετικά με τη βία αλλά και για την άποψή τους σχετικά με το πώς ε, ε, βίωσαν τα διάφορα μέτρα που ήδη έχουν θεσπιστεί στα κράτη-μέλη. Θα τοποθετηθούν λοιπόν αυτές οι γυναίκες και νομίζω ότι οι απαντήσεις τους ε, θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική δράση μας. Άλλοι μίλησαν για τις ε, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και για τα κέντρα υποδοχής των θυμάτων. Πραγματικά πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων Λοιπόν, αυτές οι οργανώσεις εθελοντών ε, επίσης θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη από ολόκληρη την κοινωνία. Δεν μπορούμε δηλαδή να ε, αναμένουμε να υπομισθούν όλες τις ευθύνες αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να τους αναθέσουμε να σώσουν τη ζωή των ε, εκτεθειμένων γυναικών. Όλοι θα πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας, ολόκληρη η κοινωνία. Επίσης, μιλήσαμε για τη βία που υφίστανται οι ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, φιλομεταβατικοί, τρανσεξουαλικοί. Ε, προφανώς θα πρέπει να καλύψουμε και αυτό το θέμα. Κάποιος ρώτησε για ποιο λόγο αποσύρουν τις καταγγελίες τους οι γυναίκες. Μα ακριβώς επειδή αποσύρουν τις ε, καταγγελίες τους προτείνω εγώ να διώκεται αυτεπαγγέλτος το αδίκημα, να μην βασιζόμαστε στην καταγγελία των ε, γυναικών γιατί όταν ε, δέχεται, υφίσταται άλλες απειλές ε, ή ε, περαιτέρω βία οι γυναίκες, ορισμένες φορές αποσύρουν τις καταγγελίες τους ε, και δεν θα, θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Σας είπα ότι χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, την αξιοπρέπειά τους, την ακαιρεότητά τους αυτές οι γυναίκες, κυρίως όταν τελούν επαπειλούμενες, οπότε είναι σημαντικό η ολόκληρη κοινωνία να αναλάβει την ευθύνη της, να χαρακτηρίσει αυτή αυτή την πράξη ως αξιόπινη πράξη και η κοινωνία αυτεπαγγέλτος επομίζεται την ευθύνη της δίωξης. προσβλέπω ε, στην συνεργασία με τους συναδέλφους ε, ούτως ώστε να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία ε, μέσα στην έκθεσή μου. Αυτό ήδη έγινε με το πρώτο σχέδιο της έκθεσης. Ε, θα δείξω ανοιχτό πνεύμα και προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους γιατί κανείς ε, ε, από μας δεν έχει από μόνος του όλες τις απαντήσεις. Από κοινού θα καταλήξουμε στις βέλτιστες δυνατές προτάσεις. Μόνο μέσα από την συνεργασία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατά πορίσματα και προτάσεις. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την σημερινή ε, συζήτηση για αυτό το θέμα που μου είναι τόσο προσφυλές. Ε, Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Για την υποβολή τροπολογιών ε, θέτουμε την 8η Δεκεμβρίου στις 12 την καταληκτική ημερομηνία, 8 Δεκεμβρίου ε, για, ε, στις 12 για να υποβάλλετε τροπολογίες. Για την έκθεση κυρία Βένσον, στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 26 και 27 Ιανουαρίου του 2011 και κανονικά θα περάσει από την Ολομέλεια το Μάρτιο το 2011 η έκθεση. Σας ευχαριστώ και ε, θα επιστρέψω τον ε, Προεδρικό Θόκο στην κυρία Σφένσον. Eh, Ας προχωρήσουμε τώρα, πάμε στο σημείο 8, απαλλαγή για το 2009 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήμα 3 Επιτροπή. Θα ήθελα να σας θυμίσω μόνο πως ε, οι συντονιστές αποφάσισαν λόγω της, ε, του ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ε, αποφάσισαν ε, οι συντονιστές να πούν στην κυρία Γκαρσία Περέσα που είναι αρμόδια για τα θέματα προϋπολογισμού να εξετάσει αυτή την έκθεση να δούμε μήπως πρέπει να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για την απαλλαγή 2009 και χαιρόμαστε που η κυρία ε, Γκαρσία Πέρες δέχτηκε να αναλάβει και αυτό το θέμα. Ε, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Μια και ο χρόνος αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει και σε σχέση και με τις παρουσίες των συναδέλφων αυτό το απαιτείται να είμαι σύντομη. Αυτό σε σχέση με την νομοδότηση αυτή είναι κάτι το οποίο είχαμε μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι σημαντικό το εγχείρημα και έχει νόημα. Κυρίως πρέπει να εμείνουμε και να επιμείνουμε σε δύο θέματα. Αρκετές φορές κάναμε λόγο για την ανάγκη του mainstreaming, της εξίσωσης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, υπό την προοπτική της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θέσει και έχουμε ζητήσει να είναι σεβαστό και στο ελεκτικό συνέδριο και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση, προαγωγή της ισότητας ως θεμελιώδους αρχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει λοιπόν τις πρωτοβουλίες της σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι πτυχές ισότητας των φύλων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις φάσεις της δημοσιονομικής εργασίας του προϋπολογισμού, την κατάρτιση, την συγκρότηση και την, ε, τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Και σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που θετικά ε, λαμβάνουμε υπόψη, αναφέρονται δράσεις υπέρ των γυναικών χρηματοδοτημένες υπέρ από το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει πέρα από αυτό να γίνουν και άλλες εκθέσεις για την εφαρμογή και λήψη συγκεκριμένων μέτρων της προώθησης της ισότητας των φύλων με βάση τις ε, ε, ε, πρωτοβουλίες και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που θα αξιολογούν την πτυχή της ισότητας των φύλων σε συγκεκριμένες δράσεις. Επιπλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα μελλοντικά λειτουργικά προγράμματα θα πρέπει να γίνονται υπό την ανάλυση της αγοράς εργασίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια διαδικασία επιλογής προγραμμάτων που θα είναι επαρκή υπέρ της ισότητας κατάρτιση, παιδεία, εκπαίδευση για τις γυναίκες στα κράτη-μέλη και στα λειτουργικά προγράμματα να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες σε κάθε μια από ε, τις πτυχές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Διαφορετικά εκείνο που θα κάνουμε θα είναι, θα δρομολογούνται πρωτοβουλίες που δεν θα αντανακλούν την ίδια την πραγματικότητα και την ένταξη της ε, γυναίκας στην αγορά εργασίας. Δεν θα ανταποκρίνονται οι ανάγκες με, τις, ε, με την πραγματική ζήτηση και πρέπει στην έκθεση αυτή να το λάβουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου για τα χρεωστήτως καταβληθέντα στο πρόγραμμα Δάφνη. Θα πρέπει να αναζητηθεί και να διευκρινιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί επαρκής εκτέλεση του προγράμματος στο μέλλον. Το πρόγραμμα Δάφνη για αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι θεμελιώδου σημασία θέμα. Κάναμε λόγο μόλις για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να δρομολογηθούν υπέρ της ε, καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών. Κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Είναι η Δάφνη ένα θεμελιώδες πρόγραμμα ως πρωτοβουλία και πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το ότι γίνεται ανεπαρκής χρήση αυτής της πρωτοβουλίας. Παρόλα αυτά όμως είναι αποτελεσματικό αυτό το εγχείρημα και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτηρήσει, να υποπτεύσει την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού του προγράμματος ώστε να υλοποιήσει τους στόχους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί και να επανέλθω να εμείνω και να επιμείνω στο θέμα της σημασίας, της σπουδαιότητας που έχει όταν ε, έχουμε ένα προϋπολογισμό να μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη την πτυχή της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις συνιστώσεις και όχι μόνο στην τελική φάση αξιολόγησης αλλά επίσης όταν κάνουμε λόγο για τις αρχικές φάσεις και την προκαταρκτική δράση η πτυχή της ισότητας των φύλων να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία Πέρες. Ε, πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα που εγείρατε. Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα της ισότητας των δύο φίλων και για τον προϋπολογισμό και πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Είναι εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Χωρίς μικρόφωνο. Μάικ. Sorry. Yes, I would like to thank... Συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρθία Πέρετ για το σχέδιο γνωμοδότησης για τη χορήγηση απαλλαγής. Στο πρώτο σημείο, το ε, κατάρτιση προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων gender budgeting. Είναι φυσικά σπουδαίο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς προϋπολογισμούς για αναφύλο ή ότι ε, περισσότερα κονδύλια πρέπει να δαπανώνται ε, σχετικά. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση, απαιτεί περισσότερο καλύτερο προγραμματισμό όσον αφορά και τον συντονισμό του των διαφορετικών τομέων και να αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της ισότητας των φύλων για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της ε, κατάθεσης του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα, gender budgeting. Υπάρχει follow-up συνέχεια που δίνεται και παρακολούθηση σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα στην ε, ανακοίνωση για την προετοιμασία, την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού αναοικονομικό έτος, προβλέποντας την ένταξη της ε, συνιστώσας της ισότητας των φύλων. Επίσης ε, μεριμνούμε και λαμβάνουμε υπόψη την ένταξη αυτού του στοιχείου όταν γίνεται και ε, εξέταση των οικονομικών, auditing, έλεγχος, εγώ είμαι ε, ελεγκτής, ελέγχουμε και ελέγχεται επίσης αν οι ίσες ευκαιρίες, η αρχή των ίσων ευκαιριών εφαρμόζεται κατά την επιλεξιμότητα και την επιλογή των ε, προγραμμάτων και σχεδίων. Τώρα, των λεχθέντων, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την επαγγελματική κατάτηση και σχετικά θέματα επιμόρφωσης. Λαμβάνουμε υπόψη, έχουμε συνειδητοποιήσει τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε και να δώσουμε συνέχεια σε μια προσέγγιση στην καλύτερη ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας και την επαρκή επιλογή εποφελουμένων ε, επιλεγόμενων σε σχέση με τα προγράμματα. Φυσικά βρισκόμαστε σε επιμερισμένη διαχείριση, shared management και η κύρια ευθύνη για τις ε, αρχές επιλεξιμότητας είναι στα κράτη-μέλη. Φυσικά προσπαθούμε να δώσουμε προσανατολισμούς και να καθοδηγήσουμε τα κράτη-μέλη και να τα συνδράμουμε παρακολουθώντας και επιτηρώντας τις ε, πρωτοβουλίες και τις δράσεις για να υπάρχουν ε, καλύτερα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία θα επιλέγονται. Ευχαριστώ κυρία Γκαρθία Πέρετ, πολύ σύντομα, απλά και μόνο για να πω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορείτε να είσαστε ήσυχοι ότι η Επιτροπή Ισότητα των Φύλων γνωρίζει ότι το mainstreaming είναι ότι η κατανομή αυτού του προπολογισμού θα είναι προ όφελο τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η πεμπτουσία, η, η κυριότερη αρχή. Και εγώ δεν είμαι επαείων σε θέματα δημοσιονομικά Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, τα στελέχη της γραμματείας της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής που με βοήθησαν εκπονώντας αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι 18 Δεκεμβρίου και κατόπιν ε, στις 26-27 Ιανουαρίου 2011 θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και το Μάρτιο, 28 Μαρτίου, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην καθήλια Αρμόδια Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και περνούμε στο σημείο 9 της Μέσης διάταξης. Καλώς ήρθατε κυρία Φιώνα Χαλ στην Επιτροπή μας. Θα μας ενημερώσετε για την ένταξη της ισότητας Τητα των φίλων στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση εκλογών. Ε, η κυρία Φιώνα Χολ διορίστηκε από την ομάδα παρακολούθησης εκλογών του Κοινοβουλίου ως αρμόδια για την εκπόνηση έκθεσης για αυτό το θέμα και για την εκπόνηση συμπερασμάτων για αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσετε σήμερα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε το απόγευμα αυτό να παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Είναι μια έκθεση για την ισότητα των φύλων και την ε, ένταξη, του, ε, ε, ένταξη αυτής της πτυχής στις δραστηριότητες όσον αφορά επιλογές και εκλογές. Δύο πτυχές θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, το θέμα της προοπτικής υπό την ευρωπαϊκή προοπτική και εκείνους που εμπλέκονται όσον αφορά θέματα εκλογών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε και το θέμα της, της εκπροσώπησης γυναικών στα κράτη-μέλη επίσης. Ξεκινώ με τα καλά μαντάτα. Όσον αφορά τη δουλειά, το έργο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Συνιστόσα έχουμε πολύ καλά στατιστικά στοιχεία για την εμπλοκή των γυναικών στην παρατήρηση εκλογών. Το 2000-2009 σε αυτά τα πλαίσια 30% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Και αν δούμε την εμπλοκή των γυναικών στο έργο όσον αφορά την ενημέρωση και τις εκλογές βρίσκεται σε αντιστοιχεία με αυτό το γενικό ε, ποσοστό είτε αν ήταν παρατηρητές ε, ως ε, ευρωβουλευτές σε μια αντιπροσωπεία, ήταν, είτε αν ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας, είτε αν ήταν επικεφαλής ε, παρατηρητές που είχαν διοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την, επι, την Επιτροπή που ήταν αρμόδια για την παρατήρηση και παρακολούθηση εκλογών από την αρχή ως το τέλος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η πτυχή της ε, εμπλοκής γυναικών σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί σε εκείνο της εκπροσώπησης των γυναικών ως Ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο και για εκείνους που εργάζονται όσον αφορά τις αποστολές ε, ε, παρατηρητών εκλογών, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα από πλευράς Επιτροπής. Πολλές φορές σε αυτές τις αποστολές και το, ίδια, το είδα η ίδια, περίπου το μισό των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, το ίμιση. Είναι ένα λοιπόν θετικό ε, μήνυμα αυτό, καλό μαντάτο όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσώπησης γυναικών. Αν δούμε όμως τον ρόλο των γυναικών, όπως παρατηρείται στις χώρες ε, και τις, ε, την, την εποπτεία εκλογών, τότε η εκπροσώπηση σε σχέση με τις χώρες δεν είναι πολύ καλή για μια συστηματική αξιολόγηση πρόσφατα των γυναικών και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται σε δύο επίπεδα. Όταν πάνε παρατηρητές σε μια ημέρα εκλογών να παρακολουθήσουν το τι συμβαίνει και όταν πάνε με ένα κατάλογο θεμάτων που πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με τις ε, κάλπες εκλογικούς καταλόγους κτλ. Σε αυτόν τον ε, στερεότυπο κατάλογο υπάρχουν ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται για το ρόλο των γυναικών στο, στα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα σε πόσα από αυτά τα εκλογικά κέντρα βρίσκονται γυναίκες που είναι παρούσες, ποιος είναι ο ρόλος τους κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, πολλές φορές έχουμε εκατοντάδες ε, τέτοια στοιχεία για την ε, συμμετοχή αυτή και με βάση αυτά έχουμε την εικόνα που αποκομίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξετάζοντας το συνολικό πλαίσιο της διεξαγωγής των εκλογών, την πολιτική κατάσταση σε μια ε, συγκεκριμένη δεδομένη χώρα, Επίσης κάνουμε μια ανάλυση των επιπτώσεων και των ε, αποστολών και των ε, εκθέσεων που συντάσσονται στο τέλος τέλος από αυτές τις επιτροπές εποπτείας εκλογών και για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες και στα κοινοβούλια κτλ. Και εδώ το μήνυμα είναι πολύ πιο ανάμεικτο θα έλεγα. Όσον αφορά τα εκλογικά κέντρα έχω δει πολλές βελτιώσεις ακόμα και σε χώρες που εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την εμπλοκή γυναικών στην πολιτική ζωή γενικότερα και συχνά υπάρχει ένα σχετικό καλό θα έλεγα επίπεδο επιδόσεων ε, όσον αφορά τις γυναίκες σε αυτό το σημείο στα εκλογικά κέντρα αν δούμε όμως την εμπλοκή των γυναικών στη συνολική πολιτική διεργασία και στις διαδικασίες συνολικά, τότε εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική. Γενικά συμφωνείτε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι ένα τρίτο των ε, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων για να μπορούν να έχουν την ε, κριτική μάζα, την κρίσιμη μάζα, ώστε να ακούγεται η φωνή των γυναικών αποτελεσματικά στα κοινοβούλια. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων δείχνουν όμως ότι αυτό πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είμαστε τέλειοι εμείς και στην Ευρώπη εμείς οι ίδιοι. Πόρο απέχουμε από την τελειότητα. Και αν δούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα συμμετοχής γυναικών στην Σουηδία 40%, Ολλανδία 41%, Φινλανδία 40%. Έχουμε όμως και πολύ αρνητικές, ε, πολύ αρνητικές επιδόσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο π.χ. από το οποίο προέρχομαι 22% συμμετοχή γυναικών. Και είναι δύσκολα τα πράγματα όταν καταλήγουμε στο να συντάξουμε, να καταρτήσουμε κάποια συμπεράσματα με ε, κάθετο τρόπο, λέγοντα τούτο ή το άλλο πρέπει να γίνει, διότι δεν έχουμε επιλύσει τα προβλήματα στην Ευρώπη όπω θα έπρεπε. Δεν έχουμε θέσει εντάξει τα του οίκου μας. Θα έλεγα σε σχέση με την επιλογή, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αυτά τα ερωτήματα. Και όχι απλά και μόνο να βάζουμε στα βρουδάκια στου καταλόγου, αλλά σε συζήτηση με τα μέλη κυβερνήσεων και όταν καταλήγουμε σε τέτοιες συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αυτά τα ερωτήματα. Διότι αυτό που σημαίνει καμιά φορά είναι ότι υπάρχει κάποια κρίση σε κάποιες εκλογικές πτυχές που παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο τέλος τέλος και όλοι επικεντρώνουν την προσοχή τους μόνο σε αυτό και θεωρούν ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να διατυπώνονται ερωτήσεις για τον ρόλο των γυναικών ή ε, να διατυπώνονται θέματα τα οποία αφορούν τις γυναίκες ενώ υποτίθεται θα έπρεπε να επικεντρώνουν όλη την προσοχή τους στα, σε εισαγωγικά μόνα σοβαρά θέματα που είναι εκείνα της επικαιρότητα. Πρέπει λοιπόν να, μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αυτά τα ερωτήματα και να τονίζουμε τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή και στην πολιτική γενικότερα στις χώρες αυτές και να αναγνωρίζετε και να ε, γίνεται αυτό ε, δεκτό. Είναι ένα θέμα που για μας θεωρούμε ότι ε, αφορά όλους και θα πρέπει στην πολιτική αυτή ζωή να λαμβάνεται υπόψη όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διεξοδική η παρουσίασή σας και είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα. Είναι θέματα δημοκρατίας, Και επίσης είναι θέμα επιμερισμού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι μπορούμε ενδεχομένως να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα και στη δική μας την πλευρά, στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να βελτιώσουμε τα ενίκο ούτως ώστε να έχουμε και αυξημένη επιρροή σε άλλες χώρες. Εδώ έχω τη σύνθεση μπροστά μου και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα πρότεινα να μοιραστεί το έγγραφο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα για την Επιτροπή μας. Πρέπει να δούμε αφενός πώς έχει η κατάσταση, αφετέρου έχουμε και τη σύνοψη ε, και τα μέτρα που ενδεχομένως θα αναλυφθούν. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν και για τη σημερινή παρουσίαση και για το υλικό που μας δώσατε. Μπορούμε να το ε, επανεξετάσουμε στην Επιτροπή μας ε, σε επόμενη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε. Ε, κυρία Μογά, έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ναι, ναι, ε, ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο θα κάνω, διότι θίξατε ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι προ συμφέρον μα να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί για αυτό το ζήτημα, δηλαδή η θέση των γυναικών μέσα στις πολιτικές ομάδες η δημοκρατία, ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας και οι θέσεις που κατέχουν οι γυναίκες ε, στις δημοκρατικές ε, διαδικασίες ε, είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και θέσεις που κατέχουν οι γυναίκες στις πολιτικές ομάδες. Με πυγμή και αποφασιστικότητα θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το τομέα. Κυρία Χολ. Πράγματι και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητάμε όταν συναντιόμαστε με τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή ποια μέτρα λαμβάνουν για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες τι είδους υποψήφιες βάζουν στις εκλογές γιατί είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ε, αρκετοί υποψήφοι ε, είναι προφανές ότι θα εκλεγούν κιόλα αρκετοί. Ε, τα μέτρα λοιπόν τα οποία λαμβάνονται επικύλουν σε ορισμένες χώρες. Βλέπουμε ότι έχουμε συγκεκριμένες ποσοστώσεις για τις γυναίκες, σε άλλες πάλι ποσοστώσεις υπάρχει μια μικρή ενθάρρυνση να υπάρχει και εκεί μια ποσόστοση, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς τα χρήματα που χρειάζονται για να ε, μπει ως υποψήφιος. Όταν λοιπόν μιλάμε για πολιτικά κόμματα, πρέπει πράγματι να ληφθούν ε, θετικά μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή. Και εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα. Μερικές φορές υπάρχουν κάποια μέτρα για, τα, για τις ποσοστώσεις ε, των γυναικών ε, και παρόλα αυτά οι γυναίκες ε, παρακάμπτονται με το να μην μπαίνουν ε, επικεφαλής ε, καταλόγων της λίστας ή να μην προβάλλονται επαρκώς. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε κυρία Χόλ και έτσι ολοκληρώνουμε και την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 ε, με ψηφοφορίες και έχουμε κάνει και διάφορες αλλαγές ε, στην ημερήσια διάταξη. Πάντως για τη σημερινή συνεδρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και ευγενικά ευχαριστεί η και τους διερμηνείς. Ε, εσάβριον στις 9. Ευχαριστώ πάντως για σήμερα.